A ver, eh, Tenemos ya nuestra directora general Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά το γεγονό ότι έχουμε πολύ λίγου συνάδελφου στην αίθουσα, θα αρχίσουμε τη μερίσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα, σημείο Α, πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό, θέλω να σας πω ότι τα Ιταλικά, για λόγους τεχνικούς, επειδή έχουμε την οθόνη πίσω μας, κάθεται στην καμπίνα αριθμός 4. 5, όχι. 5 λέει πρόεδρο μου, είπαν 5, έφυγε από το 4 και πήγε στο σημείο 5. Στο 5 λοιπόν, για να ακούσετε τα Ιταλικά 5. Λοιπόν, όπως πάντα θα πω τα εξή. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται απευθείας από το ίντερνετ του Κοινοβουλίου Έχουμε πρώτα απ' όλα την ε, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 18 Οκτωβρίου. Και αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σήμερα και αύριο δεν ε, υποβληθούν παρατηρήσεις, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί. Δεύτερον, το σημείο 3. Ανακοινώσει Πρόεδρου. Απλώ θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μία αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Αλίας που αποτελούσαν η κυρία Λοβίκη, και οι κύριοι Καντέκ, Χάγκλουμ και Φερέιρα, καθώς και εγώ, πήγαμε στη Μαυριτανία για να μιλήσουμε με τις ε, αρχές και με τον κλάδο για το μέλλον των αλληλευτικών σχέσεων και να δούμε πώς αναπτύσσεται και η αλληλευτική πολιτική της Μαυριτανίας. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε συνεδριάσει σε πολλά επίπεδα, συναντήσαμε και τον ε, Πρωθυπουργό, και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με εκπροσώπους ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν θα μακρηγορήσουμε, δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα σας υποβάλουμε μία έκθεση πιο λεπτομερή που θα σας παρουσιάσουμε την επόμενη φορά. Ε, δυστυχώς, δεν ε, μπορέσαμε να κάνουμε ταξίδι στο Βαριμπού, δεν ε, έχουν ακόμη διευκρινηθεί οι αιτήσεις, αλλά μέσα στη Μαυριτανία περάσαμε ωραία. Επίσης, πρέπει να σας πω, αιτήσει πολλών συναδέλφων. Συναδέλφων. Άλλων που έρχονται πολλές φορές. Και άλλων όπως ο κύριος Ντέβις που δεν έρχεται πολύ συχνά μου ζήτησαν να δείξουμε ένα ντοκιμαντέρ για τον κόκκινο τόνο όπως μου είχε ζητηθεί, δεν δέχτηκα να δούμε το ντοκιμαντέρ αυτό πριν, αλλά στο τέλος συνεδρίας, για δεδομένου ότι θα πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να πει οι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα και έτσι θα ενημερωθείτε και με αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, περνούμε τώρα στο σημείο 4. Ανταλλαγή απόψεων με την Lowry Evans, Γενική Διευθύντρια της Γενική Διεύθυνση Θαλάσσια Πολιτική και Αλία σχετικά με την παρουσία του προγράμματο εργασία Γενική Διεύθυνση Θαλάσσια Πολιτική και Αλία 2011 και τα πορίσματα του Συμβουλίου Αλία τη 26η Οκτωβρίου. Και όπω ξέρετε, ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έντονη συζήτηση που έγινε σε πολλά σημεία. Η κυρία Γενική Διευθύντρια έρχεται ετήσι της για πρώτη φορά στην ε, συναντήσή μας. Ορίστηκε πολύ πρόσφατα ως διευθύντρια. Την ευχαριστώ που ζήτησε να μας δει. Εγώ βεβαίως την έχω συναντήσει αρκετές ε, φορές και εκτός συνεδριάσεων κομισιών. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλό να έρθει εδώ η κυρία Γενική Διευθύντρια για να τη γνωρίσετε. Και πρέπει να σας πω ότι το λίγο χρόνο που ασκεί τα καθήκοντά της διαπίστωσα ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στον αλλιευτικό τομέα. Και όταν ορίστηκε ως Γενική Διευθύντρια, διαπίστωσα αρκετά σύντομα ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους σχετικούς φακέλους και γνωρίζει όντως πάρα πολύ καλά την κοινή αλλιευτική πολιτική, πράγμα πολύ θετικό τη σήμερα ημέρα. Της δίδω αμέσω το λόγο και μετά Θα κάνουμε ανταλλαγές απόψεων, θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές. Το λέγω έτσι χωρίς να βλέπω και μεγάλη παρουσία συντονιστών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ήβαν, σας δίνω λοιπόν αμέσω το λόγο και σας καλωσορίζω. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, πολύ χαίρομαι που έρχομαι για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβα πρόσφατα Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλίας. Είμαι στη φάση της μάθησης τώρα και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω αυτά που θα, μας, θα, θα μου πείτε. Από τον Ιούλιο έγιναν διμερείς επαφές και ανταλλαγές απόψεων όπως ακούσαμε σχετικά με τα πιο ενδιαφέροντα για σας θέματα και πρέπει ευθύς εξ αρχής να σας πω ότι προσβλέπω στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να ε, μιλήσουμε θα είμαι έτοιμη. Παρακολουθούσα ήδη με μεγάλο ενδιαφέρον και του σύνεγγυ τη συνεδριάσει, σα και είναι προφανέ ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα μα ε, δίνει μια νέα πρόκληση στι εργασίε μα. Με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατά το παρελθόν. Μπορούμε λοιπόν να βράξουμε την ευκαιρία τις κοινοτικέ πολιτικές ή τις ενωσιακές πολιτικές να τις φέρουμε πιο κοντά στους πολίτες. Εγώ αναλαμβάνω τη δέσμευση να συνεργαστώ για να γίνει αυτό. Μαζί να το καταφέρομαι στην κοινή πολιτική ελίας. Γιατί, για να το πούμε καθαρά, αν δεν γίνουν σημαντικές οι πολιτικές μας για αυτά που θέλουν να κάνουμε οι πολίτες, τότε ε, δεν ε, θα έχουμε αποτέλεσμα. Θα σας παρουσιάσω καταρχήν την έκβαση του Συνόδου του Οκτωβρίου, 26 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο και τις βασικές γραμμές του προγράμματος εργασίας μας για τον επόμενο χρόνο. Αρχίζω με το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Γενικά η Κομισιόν είναι ευτυχής από την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αλλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική ήταν ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση, πρέπει να πω, από, μέσα από το πρίσμα της, Κομισιόν. Πρέπει να πω ότι υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία και δουλέψαμε καλά και με τα κράτη-μέλη. Για πρώτη φορά θέλω να καταλάβετε ότι από τη δική μας την πλευρά ε, ε, επετέχθη ένα συνεκτικό αποτέλεσμα το οποίο σέβεται τη δέσμευση για το MSY, δηλαδή την ε, μέγιστη απόδοση, διατηρήσιμη απόδοση και μείωση της θνησιμότητας όλων των αποθεμάτων των ψαριών. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Κομισιόν Θέλαμε να προσπαθήσουμε να δούμε. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε απλά πλαίσια ε, μια γραμμή πλεύσης στο Συμβούλιο που θα είναι καλή και από άποψη οικονομική και από άποψη οικονομική για τον κλάδο. Όμως είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και για τη Σαρδελόρεγκα, το ΣΠΡΑΤ, που είναι πολύ σημαντικό για τη βαλτική αλία και τη μεταποιητική βιομηχανία σε αυτές τις χώρες. Η Επίτροπος Δαμανάκη για την Κομισιόν ε, μίλησε για την μεγάλη ανάγκη μείωσης της θνησιμότητας. Ε, ήταν πολύ σημαντικό αυτό και για την Σαρδελόρεγγα. Αλλά αυτό δεν συμπεριελήφθη. Η γραμμή πλεύσης της Επιτρόπου Δαμανάκη για την Κομισιόν είναι ότι οι αποφάσεις για τα ΤΑΚ θα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά πορίσματα και να είναι συμβατά με τα πολιετή υφιστάμενα προγράμματα για τον έλεγχο. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του τομέα της αλίας και να αποφύγουμε την κατάρρευση των αποθεμάτων με καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν τότε. Οι, τα βασικά, οι βασικές πτυχές της ομόφωνης συμφωνίας στο Συμβούλιο είναι οι εξής. Υπήρξε κοινή δήλωση Συμβουλίου Κομισιών για την ανάγκη να υπάρξουν σχέδια διαχείρισης ε, για τα πελάγια είδη για, το, για την επίτευξη του στόχου του, της μέγιστης διατηρήσιμης απόφασης μέχρι το 2015. Αυτό θα ισχύει και σε άλλες περιοχές, αργότερα και για άλλα είδη. Υπήρξε αποδοχή ότι η τεκμηριωμένη αλληλεία ε, για τα αλληλεύματα μειώνουν τις απορρίψεις. Αυτό θα το δούμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Ε, ο κύριος Στίβενσον ε, το γνωρίζει αυτό. Για τα αποθέματα, οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής. Ο τίτλος είναι «Μείωση κατά 30% για το ΤΑΚ της ε, Δυτικής Ρέγκας» και θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό το ΤΑΚ τον Δεκέμβρη όταν θα αποφασίσουμε για το ΤΑΚ στο Σκαγεράκι Κατεγάτη στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την Νορβηγία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με περικοπή αλληλευτικών ε, δυνατοτήτων και είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για τους ενδιαφερομένους αλληλείς. Κατέστη ε, αναγκαίο να γίνει πρόταση και να υπάρξει συμφωνία γιατί τα αποθέματα είναι σε κακή κατάσταση. Και μάλιστα αυτό ήταν κάτι που όλα τα κράτη-μέλη ε, είχαν ξεκαθαρίσει ως μοναδική διέξοδο και εναλλακτική. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι για κάποια αποθέματα σημειώθηκε αύξηση στα τάκ, δηλαδή συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Ε, το ανατολικό ανέβηκε κατά 15% για το μπακαλιάρο και το δυτικό κατά 16%. Ε, το δίδαγμα από εδώ είναι ότι τα προγράμματα διαχείρισης όπου υφίστανται και εφαρμόζονται σωστά δίνουν καλύτερα αποτελέσματα για τα αποθέματα και ανοίγουν καλύτερες ελευτικέ δυνατότητες για τους αλληλείς. Έτσι αποκρισταλώθηκαν οι παλιές αποφάσεις για τη διαχείριση που πέρασαν ως οικονομικά ε, ωφέλη για τον τομέα. Η μείωση του 24% για τη Σαρδελόρεγγα που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχτεί η Κομισιόν. Δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε, διότι ακόμα και αν αυτό μεταφράζεται σε καμία αύξηση της θνησιμότητας ε, του αποθέματος, σημαίνει ότι δεν επιτελείται πρόοδος σε σχέση με το στόχο του 2015 για το MSY. Και αυτό ε, την ενδιαφέρει πάρα πολύ την Κομισιόν να το πετύχει. Το Συμβούλιο επίση έκανε ανταλλαγή απόψεων για τι ετήσιε διαπραγματεύσει που επίκυνται τώρα με την Νορβηγία. Φέτο οι διαπραγματεύσει θα είναι δύσκολε γιατί, ο ο, ε, γιατί το μπλε γάδος που ενδιαφέρει πολύ είναι σε κακή κατάσταση και μάλιστα από την άλλη πλευρά η Νορβηγία προσφέρει ε, 12% παραπάνω στον αρκτικό τόνο, ε, γάδο, συγγνώμη. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ε, η οποία αποτελεί ένα δίλημα για τα κράτη-μέλη, έτσι όπως το παρουσιάσαμε. Και ένα άλλο ζήτημα που το ξέρει πολύ καλά η Επιτροπή σας, είναι το πρόβλημα που έχουμε το σκουμπρί με την Ισλανδία και τις Φερόες. Αυτό είναι ένας άλλος παράγων που περιπλέκει τα πράγματα. Οπότε Λάβαμε υπόψη μας ε, τις ανησυχίες και απόψεις των κρατών μελών και θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Ο στόχος εδώ είναι να έχουμε μια ισόρροπη συμφωνία με την Νορβηγία εξ ονόματος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί ε, θα το δουν αυτό στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Είμαι βεβαία ότι γνωρίζετε ήδη πολύ καλά ότι είχαν οι Υπουργοί ανταλλαγή απόψεων για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ICAT. Οπότε ε, διαβάσατε και τον τύπο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις και η δήλωση της Κομισιόν δημοσιεύτηκε στο website, οπότε δεν θα τα πω αυτά. Ε, όμως, ίσως υπάρχει κάποια παρεξήγηση η Κομισιόν. Δεν έθεσε πρόταση επιτάπητος για τάκ 6.000 τόνους για το κόκκινο γάδο. Αυτό που ήθελε είναι να προβληματιστεί με τα κράτη-μέλη σχετικά με το πώς θα επιτύχουμε τους στόχους μας για την αναδημιουργία του αποθέματος του κόκκινου τόνου, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να, μέχρι το 2020 να έχουμε τη θαλάσσια στρατηγική για τους στόχους της υλοποιημένους. Η Κομισιόν είπε λοιπόν ότι η σημαντική μείωση του ΤΑΚ θα πρέπει να εξεταστεί, χωρίς όμως να γράψει κανένα νούμερο στην πρόταση. Ε, σίγουρα γνωρίζετε τις αντιδράσεις πολλών κρατών μελών που ζητούν μια μετακύληση των 13.500 τωρινο τορινό είναι αυτό. Άλλα κράτη-μέλη δεν έβαλαν νούμερα, αλλά υπογράμμισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του αποθέματος επί τη βάση της αρχής της προφύλαξης και τα επιστημονικά δεδομένα. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε ε, μέτρα που και πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και να έχουμε και συνέπεια σε αυτά που λέμε στα διεθνή φόρα. Αύριο θα παρουσιάσει η Κομισιόν στο Συμβούλιο μια πρόταση για διαπραγματευτική εντολή για την επόμενη σύνοδο του ICAT και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για το περιεχόμενο της πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας συμφωνίας πλαίσιο. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, οι Υπουργοί συζήτησαν τα αποτελέσματα της ε, διεθνούς διαπραγμάτευσης ε, που έγινε το Σεπτέμβριο στο Χάλιφαξ. Είναι κρίμα πραγματικά που οι συζητήσεις στο Συμβούλιο επικεντρώθηκαν κυρίως ε, σε θεσμικά θέματα σχετικά με την διαπραγμάτευση και τη διεξαγωγή της και όχι τόσο στα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα από εκεί ήταν πολύ καλά από την άποψη της διατηρησιμότητας και τα επιστημονικά δεδομένα και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό μακροπρόθεσμα για τον κλάδο. Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν για τις αυξήσεις των ΤΑΚ ε, για τα συγκεκριμένα ψάρια είναι πολύ σημαντικά για το γάδο για παράδειγμα και επίσης οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτό. Όμως ε, ε περιορίστηκε, ε, απαγορεύτηκε η αλία για γαρίδες και μειώθηκαν τα ΤΑΚ σε μια άλλη περιοχή. Αυτό είναι βραχυπρόθεσμο, αλλά όχι μακροπρόθεσμο ε, μειονέκτημα για κάποια κράτη-μέλη, Εσθονία, Λετωνία και Λιθουανία συγκεκριμένα. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασία γρήγορα για το 2011. Έγινε ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο στο Στρασβούργο πριν από λίγε μέρε και μετά η Επίτροπος υιοθέτησε, ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας. Ε, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι η στρατηγική προτεραιότητα για το 2011. Όπως σας είπα, σε κάποιους στις διμερείς μας συναντήσεις ήδη, οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση θα είναι μεγάλη πρόκληση. Θα είναι ε, σκληρές διαπραγματεύσεις. Η Κομισιόν θα χρειαστεί όλη τη βοήθεια που θα μπορέσετε να προσφέρετε ως συνομοθέτες, ούτως ώστε από κοινού να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε τη διατηρησιμότητα των ευμάτων και των αποθεμάτων. Παράλληλα θέλουμε να συμβάλλουμε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 εργαζόμενοι προς την κατεύθυνση μιας στεναρότερης οικονομικής απόδοσης χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη και συνοχή. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι ένας κλάδος αλίας που θα δίνει ε, καλύτερο εισόδημα, περισσότερες θέσεις εργασίας και θα στηρίζεται σε υγιείς οικονομικές, κοινωνικές αρχές και επιστημονικές. Έτσι η μεταρρύθμιση θα ε, έρθει σε ένα πακέτο που θα αποτελείται από πέντε μέρη. Καταρχήν θα υπάρχει μια ε, γενικότερη ανακοίνωση της Κομισιόν που θα εξηγεί το περιεχόμενο της πρότασης και θα αναδεικνύει τις ιδέες της Κομισιόν για όλους τους τομείς που δεν θα αποτελέσουν κομμάτι του νομικού μέσου ή νομοθετικού μέσου, γιατί χρειάζονται περισσότερη πρόοδο, όπως ας πούμε θέματα για το τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε τα επιστημονικά μας πορίσματα για το μέλλον. Αυτό είναι, θα είναι ένα πρώτο γενικότερο πολιτικό έγγραφο. Η βασική νομοθετική πρόταση θα είναι το βασικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ε, ούτως ώστε να αρχίσει η μεταρρύθμιση και να τεθεί σε εφαρμογή. Θα υπάρξει νομοθετική πρόταση για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στην αγορά. Θα δούμε την τομεακή οργάνωση, το ρόλο των οργανώσεων των παραγωγών για τη βελτίωση της διαχείρισης ε, όλων των θαλασσοκαλλιεργειών και το, την εμπορία των αλλιευμάτων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Επίσης θα ξαναδούμε τα μέσα που διασφαλίζουν τη σταθερότητα της αγοράς και πληροφορίες μέσα από το σύστημα επισήμανσης ε, η ετικετοθεσία που θα ενημερώνει τους ε, ενδιαφερομένους. Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τη διεθνή διάσταση της ε, κοινής αλληλευτικής πολιτικής που θα καλύπτει περιφερειακές οργανώσεις, διεθνείς οργανώσεις και τις αλληλευτικές συμφωνίες συνεργασίας. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές μας πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές και τέλος θα υποβάλουμε νομοθετική πρόταση για ένα ταμείο που θα στηρίζει την κοινή αλληλευτική πολιτική, την υδατοκαλλιέργεια και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Εδώ έχουμε υπόψη μας ε, την ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών μέσων που χρειαζόμαστε ώστε το μελλοντικό ταμείο να στηρίζει τους στόχους της ε, ε, πολιτικής αλληλεία και θα συμβάλλει στο ευρύτερο πλαίσιο που έχουμε διατυπώσει στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις, για το νέο ταμείο που προγραμματίζεται τον Ιούλιο 2011 μαζί με τις άλλες προτάσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε στο εσωτερικό μας, στο εσωτερικό μας ότι το μεταρρυθμιστικό πακέτο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Μαΐου 2011. Βεβαίω ε, θα συνοδεύεται και από μελέτη επιπτώσεων. Σα ενδιαφέρουν και οι άλλε πρωτοβουλίε του προγράμματό μα, γνωρίζω. Τώρα δουλεύουμε, για παράδειγμα, στα πολιετή προγράμματα ή σχέδια και για τον Σολομό τη Βαλτική και για τα, θαλάσσια, τα θαλασσοπούλια και για το χωροταξικό σχεδιασμό και στρατηγικές ε, και για τις ε, ε θαλάσσιες λεκάνες ε, και για τον Ατλαντικό. Δεν είμαι σε θέση να δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά πριν από το τέλος του έτους θα έχετε, είμαι βεβαία, πλήρη στοιχεία για τον προγραμματισμό μας. Σταματώ λοιπόν εδώ για να σας δώσω και χρόνο να κάνετε ερωτήσεις και να υποβάλλετε και σχόλια. Σας ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Τις εξής. Ήδη στην συνεδρίαση που είχαμε την τελευταία φορά στο Στρασβούργο με την Επίτροπο, της, είπε, της είπα κάτι και θα το επαναλάβω. Συμφωνούμε όλοι με το να ακολουθήσουμε τις επιστημονικές συστάσεις και πιστεύω ότι κανείς, ούτε εντός Συμβουλίου, ούτε εκτός, θέλει να λάβει οποιαδήποτε απόφαση που δεν βασίζεται σε συστάσεις επιστημονικές. Ξέρουμε όμως ότι έτσι προσφέρονται διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχει μόνο μία και μοναδική ερμηνεία, αν θέλετε. Είπαμε λοιπόν και εμείς ότι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αηφορία των πόρων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εναρκτικές λύσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθούμε, ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Και ξέρουμε ότι δεν ακολουθούν πάντα αυτές οι επιστημονικές συστάσεις πάντα αυτό το κριτήριο το κοινωνικό-οικονομικό. Επίσης, στις ε, περιφερειακές ε, ε, συναντήσεις που γίνονται με τους αλείς και θα το συζητήσουμε αυτό του κόκκινου τόνου. Ακούσαμε να γίνονται διάφορες παρατηρήσεις για διάφορα θεσμικά θέματα, για διάφορα θέματα συντονισμού. Και μας μας απασχολεί το θέμα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με τους συντονιστές και θα ήθελα να συναντηθώ με εσάς και με την Επίτροπο για να σας εξηγήσω ποια είναι τα θέματα τα οποία βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει και μπορούμε και δικαιούμεθα εμείς να παρακολουθούμε στα πλαίσια των διαφόρων συμβάσεων που έχουμε Δεδομένου ότι επαναλαμβάνω, αυτά είναι εξουσίες που μας δίδει πλέον η συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το θέμα το θεσμικό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Δεύτερο, θα ήθελα να πω, και το λέω εδώ δημόσια, ότι εγώ δημοσίως και εγώ πολλές φορές ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, είχα στις επισκέψεις που μου έκαναν διάφοροι εκπρόσωποι του κλάδου την εντύπωση ότι, έγινα, ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τις στρατηγικές επιλογές πολλές φορές της Επιτροπής. Εμένα λοιπόν αυτό με απασχολεί. Τα συμβαλόμενα μέρη ε, που είναι συνήθως σήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να έχουν τέτοιου είδους ανησυχίες και θα πρέπει με ορθολογισμό να εξηγούνται κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι σωστό να σας το πω αυτό. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι μου ε, έλαβα διάφορες επικριτικές επιστολές από τον κλάδο, από την Κοζέκα, από την Κόπα, στις οποίες αναφέρεται ότι τελευταία και πριν από τις συναντήσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Άλλιων δεν θεώρησε σωστό να συναντήσει εκπροσώπους του κλάδου η Κομισιόν. Το λέω αυτό διότι το ίδιο συμβαίνει και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πιστεύω ότι αυτή η έλλειψη κατανόησης ή το ότι δεν υπάρχει συζήτηση ανοιχτή για αυτού του ίσο θέμα με την κοινωνία των πολιτών είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το πούμε εμείς στην Κομισιόν, διότι εμείς ως πολιτικοί είμαστε αποδέκτες αυτών των ανησυχιών και των επικρίσεων που υποβάλλουν οι πολίτες. Τα λέγω αυτά διότι θέλω να ξέρετε ότι αυτά είναι κάποια από τα θέματα που μας απασχολούν. Τώρα όσον αφορά το θέμα το νομοθετικό. Και βλέπετε ότι δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να σα πω ότι αυτό το που είπατε ότι υπάρχουν οι δυνατότητε, ε, ότι υπήρχε δυνατότητα αλληλεία στην Βαλτική και μας είπατε ότι είναι κάτι το οποίο ομόφωνα ως απόφαση απερίφθη, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, γιατί βλέπουμε πολλές φορές, ότι όλο και δύσκολες γίνονται οι σχέσεις μεταξύ Βουλίου και Επιτροπής. Διότι εμείς βάσει του σχετικού άρθρου της συνθήκης. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλα σε θέματα, τάξη και άλλα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και το ότι υπάρχει έλλειψη κατανόησης μεταξύ ε, Συμβουλίου και Επιτροπής είναι κάτι που επίσης ανησυχεί τον κλάδο. Τώρα, για το νομοθετικό, για το πρόγραμμα. Δεν θα σας κάνω καμία παρατηρήση, αλλά θα ήθελα για τα πολυετή προγράμματά σας και αν θέλετε μου το εξηγείτε στο τέλος, το θέμα αυτό του Μερλούκιου να μου το εξηγήσετε. Μας είπατε ότι υπευλήθη μία πρόταση και απεσύρθη, αλλά δεν ξέρω, κάπου κάτι λέγεται, δεν μπορώ να το βρω, εν πάση περιπτώσει. Μας είπατε ότι κάτι άλλαξε. Ε, ποιες είναι οι προθέσεις σας αυτή τη στιγμή, θα κάνετε πρόταση για την αλία του Μερλούκιου του Βορρά ή αργότερα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, στους συντονιστές. Για το ΕΛΚΑ. Βλέπω τον συνάδελφο Κάντεκ. Θέλετε εσείς το λόγο κύριε Κάντεκ ή να δώσω άλλο συνάδελφο. Δεν είναι εδώ συντονιστής, κάντε εσείς το συντονιστή. Ρωτώ τον Αντιπρόεδρο αν θέλει ο ίδιο να υπομειστεί τον ρόλο του συντονιστού ή να κάνει ερωτήσει. Εντάξει, πολύ καλά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γενική Διευθύντρια, σας άκουσα προσεκτικά και φαντάζομαι ότι είπατε ότι τα πάντα βαίνουν αισίως. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα από τη δική σας την παρέμβαση, αν σας κατάλαβα καλά. Ήσασταν στην συνεδρία του Συμβουλίου στις 26. Τα πράγματα παρουσιάστηκαν εκεί πέρα με μια κάποια δυσκολία φαντάζομαι. Χαίρομαι πολύ πάντως που βλέπω ότι εσείς κρατάτε μια θετική στάση, αλλά εγώ δεν είμαι πεπισμένος για το ότι τα πράγματα όντως βαίνουν αισίως. Όσον αφορά το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε η πρόεδρός μας, η κυρία Φράγκα, συμφωνώ απόλυτα με τη δική της την ανάλυση. Δηλαδή, προφανώς θα πρέπει να βασιστούμε στην επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό αποτελεί και θα αποτελεί πάντα τη βάση. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανεί με αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως είπε και η πρόεδρός μας και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, την κοινωνικονομική κατάσταση και επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε περισσότερο με τον επαγγελματικό κλάδο σε σχέση με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι είναι πραγματικά κρίμα που δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και προφανώ θα πρέπει πάντα να βασιζόμαστε στην επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Μόνο αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση μα για να διατηρήσουμε την α, αλία, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και να διατηρήσουμε επίσης και τα αποθέματα. Νομίζω ότι βάσει αυτών των στόχων θα πρέπει να εργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς η Επιτροπή Αλίας και οι βουλευτές της αυτό θέλουν να πετύχουν στα πλαίσια της συναπόφασης και στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Για άλλη μια φορά, πρέπει να σας πω κυρία Γενική Διευθύντρια, ότι δεν είμαι πεπισμένος ότι τα πάντα βαίνουν αισίως. Βέβαια, θα έχετε δυνατότητα να μου απαντήσετε στο σχόλιο μου αυτό λίγο αργότερα. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Γενική Διευθύντρια για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ με τα όσα είπε η Πρόεδρος για τα ζητήματα αυτά τα οποία συζητάμε. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές που είναι όλες πάρα πολύ σημαντικές για τα θέματα που συζητάμε εδώ στην Επιτροπή Ελίας. Και θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω και με τον κύριο Καντέκα. Ο επαγγελματικό τομέα αλληλεία πλήττεται πάρα πολύ στην Ευρώπη, τόσο στη Βόρεια Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο. Το είπε αυτό ξεκάθαρο ο κύριο Καντέκ. Έχουμε σημαντικά προβλήματα με τα αποθέματα. Η βιωσιμότητα των αποθεμάτων είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει. Και πιστεύω ότι ε, καθήκον μας είναι να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κοινή αλληλευτική πολιτική. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να καταφέρουμε να καταρτήσουμε σχέδια τα οποία θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αλίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των αλλιέων, οι συνθήκες πληρωμής τους, πώς μπορούμε παράλληλα να σεβαστούμε την βιοπικιλότητα και να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του κλάδου. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα του τομέα, να καταφέρουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του επαγγελματικού κλάδου. Όσον αφορά τώρα την διαχείριση σε καθημερινή βάση, κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο σημαντικοί τομείς στους οποίους θα πρέπει να εργαστούμε. Ήδη έχουμε μια σειρά συμφωνιών διμερείς συμφωνίες όσον αφορά την αλία και όπως είπε και η πρόεδρος, υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός αποκλειστικότητας όσον αφορά τις συμφωνίες αυτές και θα έλεγα ότι πολύ συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται εκτός της διαδικασίας σύναψης συμφωνιών. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο υπονομεύει τις διατάξεις της Συνθήκης Λισαβόνας η διαχείριση των ΤΑΚ και, των, και της ελευτικής προσπάθειας είναι ζήτημα το οποίο σαφώς θα πρέπει να υπάγεται σε επιστημονική ανάλυση. Όλοι συμφωνούμε νομίζω με αυτό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής οι επιστήμονες δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το όριο των 6.000 τόνων όσον αφορά τον κόκκινο τόνο δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση από την επιστημονική κοινότητα, δεν υπάρχει μια τέτοια ένδειξη τουλάχιστον. Και νομίζω τελικά ότι πίσω από την επιλογή αυτή κρύβονται διάφορες πολιτικές προθέσεις. Όταν θα χρειαστεί λοιπόν να λάβουμε μια επίσημη απόφαση, θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ομάδες συμφερόντων και αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει με τρόπο ήρεμο. Αν αναφερθούμε στο όριο το οποίο είχε αποφασιστεί πέρυσι, στην ποσόστοση δηλαδή την οποία είχε αποφασιστεί πέρυσι, η ποσότητα αυτή τηρήθηκε θα έλεγα από τους περισσότερους εκτός από κάποιους Γάλλους αλείς. εκεί πέρα είχαμε κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω όμως αν μπορούμε να πούμε ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της περσινής ποσόστοσης στο φεστινό έτος. Όταν λοιπόν κληθούμε να σχεδιάσουμε την μελλοντική ηλεκτρική πολιτική, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερο να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να δραματίσει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Και νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ε, πολύ συχνά δεν εισακούονται πολλές αποφάσεις λαμβάνονται στο όνομα του περιβάλλοντος, στο όνομα της βιοπικιλότητας και έχω πολλές φορές την εντύπωση ότι δεν ακούμε τη φωνή των αλλιέων επαρκώς. Και η συνέπεια τελικά της τάσης μας αυτής είναι ότι ενδεχομένω να μην καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιες είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεων, των αποφάσεων μας ή τουλάχιστον ποιες είναι οι συνολικές επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων για παράδειγμα όσον αφορά την οδηγία για την αλία μικρής κλίμακος στην ε, Μεσόγειο, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επιπτώσεις, η επιρροή από την απόφαση αυτή, από την οδηγία αυτή, όσον αφορά τον κοινωνικονομικό τομέα, είναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερος, περισσότερος διάλογος. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να θίξω είναι η συνολική μεταρρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική. Αυτή δεν μπορεί να γίνει προφανώ από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται μία μακροπρόθεσμη στρατηγική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το είχε πει ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε εγκρίνει μάλιστα δύο εκθέσει. Η μία έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική τη κυρία Πατρανιέδη και έχουμε και μία άλλη οδηγία για τη βιωσιμότητα τη υδατοκαλλιέργεια. Εγώ ήμουν εισηγητή για το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που εμείς εγκρίναμε τις εκθέσεις αυτές, δεν ξέρω ακριβώ ποιες θα είναι οι προτάσεις που θα δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο. Πιστεύω πάντως ότι αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να έχουμε από τη μια μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και από την άλλη μια πολιτική για την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, οι οποίες να συνδυάζονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει το σύνολο του κλάδου. Η κυρία Λόβη, μέρος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Γενική Διευθύντρια να συγχαρώ καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή συμμετοχή που είχε στις διαπραγματεύσεις που γίνανε στο Συμβούλιο. Είναι πολύ θετικό το ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Νομίζω ότι ε, καταφέραμε να ακολουθήσουμε περισσότερο τις επιστημονικές συστάσεις για τις περισσότερες ποσοστώσεις τουλάχιστον. Όσον αφορά βέβαια το σπράτιν σαρδελορέγκα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως εμείς τα θέλαμε και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Γιατί και στην περίπτωση του Σολομού της Βαλτικής δεν έχουμε ακολουθήσει ακριβώς τις επιστημονικές ενδείξεις μειώσαμε την ποσόστοση μόνο κατά 15% σύμφωνα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιστήμονες όμως μας είχαν πει ότι θα πρέπει να είχαμε πετύχει πολύ μεγαλύτερη μείωση της ποσόστοσης για το Σολομό της Βαλτικής. Περιμένουμε λοιπόν πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει το σχέδιο διαχείρισης για το Σολομό της Βαλτικής συντομότατα, Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη για ένα τέτοιο σχέδιο και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πρότασης που θα κάνει να μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο και να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε ότι η επίπτωση κοινωνικονομικά θα είναι μικρή. Σαφώ υπάρχουν και διάφορε εναλλακτικέ τι οποίε θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Πάντω δεν πιστεύω ότι έχουμε το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να θέσουμε εν κινδύνο το σύνολο του αποθέματο αυτού. Εφόσον υπάρχει μια επιστημονική βάση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο την αρχή της πρόληψης, πιστεύω. Δεν είναι σωστό, πιστεύω, να διακινδυνεύουμε το μέλλον των αποθεμάτων μας. Μιλάμε ουσιαστικά για τα μελλοντικά μας αποθέματα αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο όφελος, ακόμα και θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ζημία στον αλληλευτικό τομέα, στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Ας προσπαθούμε να διδαχθούμε κάποια πράγματα και από το παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά, πιστά τις επιστημονικές ενδείξεις. Όσον αφορά τώρα την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική και τη μεταρρύθμισή της, πιστεύουμε ότι όντως θα πρέπει να υπάρχουν μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης για όλα τα αποθέματα και θα πρέπει και γι' αυτό να ακολουθούμε τις ε, επιστημονικές ε, ενδείξεις. Και θα πρέπει και η πολιτική ελίας προφανώς να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Χαιρετήσουμε επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα θαλάσσιας χωροταξίας. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι αναγκαίο. Ασκείται ιδιαίτερη πίεση στο θαλάσσιο περιβάλλον από διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Και βλέπουμε σιγά σιγά ότι συσσωρεύονται οι επιπτώσεις από όλη αυτή την οικονομική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε επομένω να αντιμετωπίσουμε πλέον την πολιτική ελεία σαν μια πολιτική η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική περιβάλλοντο. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντάξουμε του περιβαλλοντικού στόχου στην πολιτική ελεία. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ένα καλό περιβαλλοντικό επίπεδο σε όλες τις θάλασσες με ορίζοντα το 2020. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, αυτή τον, για αυτόν τον πολύ καλό γύρο διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και ελπίζω τα πράγματα να εξελιχθούν το ίδιο καλά και το Δεκέμβριο. Grupo, ¿cómo se llama su grupo? Bueno, ¿cómo se llame? por el grupo de los conservadores ε, está el señor Stevenson. ¿Cómo se llama? Κύριε Stevenson, εκ μέρους των συντηρητικών. Thank you. Ναι, thanks very much, Chairman, and thanks. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Διευθύντρια που είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα μια ερώτηση που αφορά τα πελάγια θέματα. Καλό είναι να έχει κανείς ε, την βοήθεια των επιστημόνων, αλλά... Πέρσι το επιτρεπόμενο τάκ ήταν πολλές χιλιάδες τόνοι. Η Ισλανδία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό έξτρα, 100 τόνους συμπληρωματικού επίσης πήρε η Ισπανία. Ο κ. Κώστα να μας πει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, ακόμη και ε, δικούς μου υπολογισμούς, ακόμη και χίλιοι τόνοι περίπου ακόμη σκουμπρί είναι κάτι το οποίο παρέμεινε και νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Πολλές φορές βλέπουμε πολλές φορές αλλιευτικά σκάφη σκοτικά τα οποία προσπαθούν But Μπλε γάδο, αλλά δεν έχουν την ε, κατάλληλη άδεια. Μπορεί η Επιτροπή, γιατί για μένα είναι δύσκολο να καταλάβω κάποιους αριθμούς. Μπορεί να μας δώσει η Επιτροπή τους αριθμούς οι οποίοι είναι σε ισχύ και ισχύουν τα τελευταία πέντε χρόνια για τα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, τα τάκ για τα πελαγικά είδη, διότι υπάρχει τρομερή σύγχυση. Γίνονται και συζητήσεις, συζητείται και το θέμα του τι κάνει η Νορβηγία, τι κάνει η Ρωσία, τι μπορούν να κάνουν. Θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε εμείς ε, τα επιτρεπόμενες ποσότητες αλλιευμάτων, τα τάκ, για να έχουμε μία σαφή ιδέα. Τώρα μας φορά το πρόγραμμα εργασίας και την ε, ολοκληρωμένη ελληνική πολιτική που ακολουθείται. Συμφωνούμε τις αρχές, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα και διαφορές με το θέμα και των διαφόρων ε, ειδών ε, ενέργειας που χρησιμοποιείται, αλλά κανένας ποτέ δεν ζήτησε την άποψη των ειδικών του κλάδου. Γίνεται λόγος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια, την παλιροϊκή ενέργεια. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά πιστεύω ότι η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι από τη βάση προς τα πάνω, ενώ τώρα κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν ζήτησε την άποψη του κλάδου, των αλλιέων, των επαγγελματιών που έχουν να πούν κάτι. Και αυτοί αλλιεύουν σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις ζώνες, πολλές φορές περισσότερο από έναν αιώνα. Επίσης, το θέμα του χωρισμού σε περιφέρειες. Περιφέρει. Πιστεύετε εσείς ότι είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας για το μέλλον. Αλλά υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλοί που αναρωτιόνται αν είναι κάτι το νόμιμο και το Συμβούλιο έχει ερωτηματικά και πολλοί στα κράτη-μέλη είναι αυτοί που είναι αντίθετοι. αν κάνουμε μια ορθολογική και λογική πολιτική περιφερειοποίηση, να ξέρετε ότι και εμεί θα σα υποστηρίξουμε. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στου υπόλοιπου συνάδελφου και στο τέλο, αν θέλετε, κύριε Γενική Διευθύντρια, να απαντήσετε συνολικά. Ο κύριο Κούν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Γενική Διευθύντρια, ευχαριστώ πολύ. Να δούμε πρώτα το πρόγραμμα εργασίας 2011. Βεβαίως η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι το βασικό θέμα. Και εσείς ε, το υποδιαιρέσατε σε πέντε μέρη, όπου βέβαια παίζει ρόλο και ένα θέμα που σίγουρα στην διάσκεψη στο Συμβούλιο Υπουργών των Υπουργών Αλληλείας τον Οκτώβριο έπαιξε ρόλο. Δηλαδή μιλάω για την βελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Θεωρώ ότι και μέσα από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια οι εμπλεκόμενοι πρέπει να δώσουν εμπειρική ε, ε, ε, γνώμη. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Ξέρουν οι άνθρωποι επιτόπου. Επίσης η μεταρρύθμιση της πολιτικής εμπορίας, η άμεση εμπορία, οι άμεσες πωλήσει παίζουν ρόλο. Λέτε για επισήμανση ή ετικετοθεσία. Είναι σημαντικό στην Ευρώπη αυτό. Είμαστε τεράστια εισαγωγική αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σήμανση και των εισαγωμένων προϊόντων ε, ψάρια και προϊόντα αλεία. Είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των καταναλωτών. Τα πολυετή προγράμματα που επίσης αναφέρατε κυρία Evans είναι αξιέπαινα οπωσδήποτε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Σολομό της Βαλτικής, αλλά είδα ότι έχετε και για τα θαλασσοπούλια πολυετή πουλιά, ίσως και για τις ε, ε ε, που μπορεί να παίζουν ε, ε, πολύ σημαντικό ρόλο γενικότερα για το θαλάσσιο σύστημα. Επίσης, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Το Συμβούλιο Αλίας, έτσι μας είπατε, με μεγάλη συμφωνία ενέκρινε τα ΤΑΚ. Παρατηρούμε όμως ότι εδώ στην Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική η Νορβηγία, ένα αλλιευτικό έθνος, παίζει μεγάλο ρόλο και τα μέλη του Συμβουλίου Αλίας δεν, πιέσαν, δεν άσκησαν πιέσεις άσκοπα, δηλαδή αυτές οι περικοπές στη Ρέγγα 30% ε, ή στη Σαρδελόρεγγα 24% περικοπή των ΤΑΚ, αυτό θα το κάνουμε μόνο αν συνεργαστεί και η Νορβηγία, αν οι διαπραγματεύσεις δηλαδή μετά καταλήξουν θετικά. Ξέρω με τη συμφωνία με την Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το τομέα σε ό,τι αφορά τη ρέγγα της Βαλτικής και στο 3α έχει 23-24 εκεί συμφώνησαν σε μια θέση 50-50 σε μια τέτοια συμφωνία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους αλληλείς στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική. Για μένα θα ήταν επίσης κάτι άλλο σημαντικό. ΤΑΚ ε, ε, να περικοπούν ε, κατά 30%. Ιδιαίτερα στη Ρέγκα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν τέτοιες ε, περικοπές αυτής της τάξης μεγέθους για να είναι διατηρήσιμα τα αποθέματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε μιλήσει και για άλλα μέτρα. Ίσως το έχετε κάνει. Μπορεί να απαντήσετε και σε αυτό το ερώτημα. Σχετικά με τα απειλούμενα ε, αποθέματα και πώς μπορούν αυτά να προστατευτούν. Γιατί τη Ρέγγα δεν υπάρχουν πολυετή προγράμματα, ούτε διαχειριστικό πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο και το έχουν προετοιμάσει οι επιστήμονες. Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο πρόγραμμα διαχείρισης και αυτών των αποθεμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Εύανς. Μπορώ να σουμάρω κάποιες απαντήσεις. Καταρχήν τα επιστημονικά δεδομένα. Λοιπόν, η επιστήμη δεν ορίζει την πολιτική, είναι μια συμβολή στην πολιτική, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είπατε κι εσείς, το λέει και η Κομισιόν. Όμως, ο μύτος, η κόκκινη κλωστή της δουλειάς της Κομισιόν ποια είναι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βελτίωση των αποθεμάτων από εδώ που είναι τώρα δεν είναι μόνο προ το συμφέρον τη αναδημιουργία των αποθεμάτων, αλλά τη αύξηση των αλλιευμάτων μα για το μέλλον. Δηλαδή είναι προ το συμφέρον του κλάδου του ίδιου. Η... Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τα επιστημονικά πορίσματα και πάντοτε παρακολουθούμε τις εξελίξεις της επιστήμης, στηρίζουμε μια προσέγγιση η οποία θα πρέπει να φροντίσει να βάλει σε καλύτερη θέση τον κλάδο στο μέλλον από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή, πιο περισσότερες βιώσιμες θέσεις στο μέλλον, ένα κλάδο με καλύτερα αμοιβόμενε θέσεις εργασία στο μέλλον από ό,τι τώρα. Αν δεν έχετε ψάρια να πιάσετε, δεν μπορεί να έχετε ε, θέσεις εργασίας, αλληλείας και μεταποίησης. Η έμφαση λοιπόν στην επιστήμη αυτό αφορά την οικονομική βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα και Φορεία. Στη τελευταία ανάλυση αυτή είναι η θέση της Κομισιόν και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και του Κοινοβουλίου. Υπογράμμισα λοιπόν ιδιαίτερα την επιστήμη σε αντιπαράθεση με... Α, εάν έκανα μια, μια ε, αντιπαράθεση μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών και επιστημονικών δεδομένων, ε, δεν τα είπα καλά, όλα αυτά πάνε μαζί. Η επιστήμη θα πρέπει να είναι αξιόπιστη στα μάτια των αλλιέων. Και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, διότι η αλής, ο κλάδος της αλίας και τα δεδομένα του κλάδου της αλίας θα πρέπει να αναλύονται και να περιλαμβάνονται. Και πολλή δουλειά μπορεί να γίνει εκεί στο μέλλον. Εμένα με ενδιαφέρουν οι εσδήποτε προτάσεις από την πλευρά σας για να το καταφέρουμε αυτό. Το επιστημονικό ζήτημα λοιπόν αφορά και ταυτίζεται αν θέλετε με τα οικονομικά ζητήματα τυχόν προτάσεις θα τις δεχτώ με μεγάλη χαρά. Τώρα, ε, ε, σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς, ίσως είμαι δηλαδή γενικόλογη και υπεραισιόδοξη σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Δεν περιορίστηκα μόνο στο θέμα των τάξεων ε, μίλησα για την Βελγική Προεδρία, η οποία επίσης υπογράμμισε την επιστημονική σημασία όλων αυτών των δεδομένων για την οικονομική βιωσιμότητα. Είμαι πεπισμένη ότι για να βγάλουμε αποτελέσματα τα οποία θα είναι βιώσιμα από οικονομική άποψη, ε, αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάθε προσπάθεια, αξίζει τον κόπο. Θα περίμενα να χαρείτε πολύ ε, από αυτή την ε, αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον. Η Βελγική Προεδρία ε, θα πρέπει να επενεθεί τουλάχιστον ως εμείς, αν όχι και περισσότερο. Τώρα, για τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Αυτό είναι μια βασική διάσταση της συνέχισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και εσείς ε, παραδοσιακά ε, ενδιαφερθήκατε για αυτά, ε, πιέσατε για τα προγράμματα για το Μερλούκιο κλπ. Θα έχουμε προγράμματα για τα πελάγια βαλτικά ήδη. Δεν έχω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά αυτό το υπόσχομαι. Η ιδέα είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα και όσο γίνεται ταχύτερα προγράμματα διαχείρισης για τα βασικά αποθέματα. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες, θα τις επεξεργαστούμε με το Κοινοβούλιο Συνομοθέτη πρόθεσμα ε, του χρόνου. Ε, αυτά θα προχωρήσουν και θα επιταχυνθούν μάλιστα οι ρυθμοί. Μια διάσταση πολύ σημαντική για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης είναι τα τελευταία αυτά να είναι και προβλέψιμα για τον κλάδο. Ε, μου κάνατε μια ε, κριτική, νομίζω ότι δεν ακολουθήσαμε για τον Σολομό της Βαλτικής στα επιστημονικά δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, ναι, καμιά φορά υπάρχουν μαρτυρίες που αποδεικνύουν ότι η Κομισιόν δεν έδωσε έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα, προσπαθώντας να βρει μια ισορροπία με τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Η Κομισιόν καταλαβαίνει τις αναγκαιότητες που υπάρχουν στον κλάδο. Πολλές φορές δηλαδή καταλαβαίνει ότι ο κλάδος δεν πρόκειται να καταπιεί, αν θέλετε, κάποια μέτρα. Πρέπει λοιπόν να εξομαλύνουμε λίγο εμείς η Κομισιόν τις προτάσεις μας. Δεν ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν απολογούμε γι' αυτό. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι με διαφορετικό τρόπο πάνω σε αυτό το θέμα, να μας το πείτε. Για να το λάβουμε υπόψη μας για του χρόνου, για παράδειγμα. Τώρα, για την κοινή αλληλευτική πολιτική, κάποια σχόλια μας δίνουν τροφή για σκέψη. Ήδη το κάνατε αυτό για την υδατοκαλλιέργεια, ε, γιατί μελετούμε πολύ προσεκτικά τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Για την περιφερειακή διάσταση, κυρία Σίμψον, ε, επίση προβληματιζόμαστε έντονα. Είμαστε ανοιχτοί ακόμα. Είμαστε ανοιχτοί για επικοδομητικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής σε κάθε θέμα, σε κάθε ε, πτυχή της. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη αυτών των διαστάσεων της πολιτικής μας από το Κοινοβούλιο. Μετά η εξωτερική διάσταση, να πω και γι' αυτό, το σχόλιο σας είναι ότι τα συμβαλόμενα μέρη ενοχλούνται από την αλλαγή της πολιτικής. Το λαμβάνω υπόψη αυτό που είπατε, το σημειώνω. Από ό,τι γνωρίζω συζητούμε με όλους τους μεγάλους διμερείς εμπορικούς εταίρους. Αν μας έχουν ξεφύγει κανένα δυο, θα καλύψουμε το κενό. Γιατί στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις στο IFMO η ιδέα είναι οι βασικοί εμπορικοί διαπραγματευτές να στοχεύουν λίγος πολύ προς την ίδια κατεύθυνση και να προσπαθούν να επηρεάσουν με ε, το σωστό τρόπο προς ε, αμοιβαίο όφελος ε, το, την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα το λάβω υπόψη μου. Ίσως ό,τι αφορά τη δουλειά του Κοινοβουλίου και το ρόλο του Κοινοβουλίου στις πολυμερείς και διμερείς συζητήσεις, μπορώ να πω αυτό που είπε η Επίτροπος Δαμανάκη ήδη, και ο αντιπρόεδρος ε, Σεύκοβιτς της Κομισιόν υπόσχομαι ότι όπως είπε και η Επίτροπος Δαμανάκη ότι θα κάνουμε το μάξιμο που μπορούμε στα πλαίσια των διοργανικών συμφωνιών το απόλυτο μέγιστο σας εγγυώμαι ότι θα υπάρξει όλη η απαραίτητη και όλη η δυνατή καλή θέληση και συνεργασία από την πλευρά μας, γιατί και προς το δικό μας το συμφέρον να είναι ενημερωμένο επί της ουσίας στο Κοινοβούλιο ε, για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει εδώ καμία ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ μας. Μου ξέφυγε κάτι? Απάντησα σε όλα. Α, για τα πελάγια ήδη. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Θα, επανέλθουμε σε σας διμερός μέσω της, και μέσω της γραμματείας, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που θα σας δώσω και στα άλλα μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να κάνω συμπληρωματικό σχόλιο σε σχέση με τις επιστημονικές συστάσεις. Απλώς και μόνο πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την αναθεώρηση του 7ου πρόγραμματος πλαισίου. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ε, συγκεκριμένο στόχο στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, πράγμα που δεν συμβαίνει στο 7ο. Και βεβαίως να δώσουμε και τα κατάλληλα κονδύλια επαρκή, περισσότερο από ό,τι έχουμε ούτως ή άλλως σήμερα, διότι υπάρχει έλλειμμα στόχων και έλλειψη κονδυλίων. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο τομέας, ακόμη και οι επιστημονικοί παραγοντέ ζητούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι γίνονται. Και όλα αυτά δεν γίνονται διότι δεν έχουμε ούτε συγκεκριμένου στόχου στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ούτε αρκετά κονδύλια. Αν θέλουμε ο προγραμμα πλαισιο ουτε αρκετα κονδυλια αν θελουμε ο στόχο μας να είναι μέχρι το 2015 όλα τα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ε, ε, να έχουν τη σωστή αξιολόγηση ανάλογα με την απόδοσή τους, θα πρέπει να ξέρουμε περί τίνους ακριβώς πρόκειται. Θα πρέπει βάσει επιστημονικών παρατηρήσεων να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι συγκεκριμένα. Άρα θα πρέπει στο επιστημονικό τομέα να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Είναι από τους στόχους τους οποίους θα πρέπει να θέσουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει, όπω σα είπα, στα πλαίσια αναφέρωση παρόντος προγράμματος και για να καθορίσουμε το επόμενο. Διότι δεν θα πρέπει να έχουμε μεγάλου ιτημένους και χαμένους και ο που να κερδίζουν από όλη την υπόθεση. Κυρία Γενική Διευθύντρια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας για την ε, παρουσία σας. Θα συνεχίσουμε να μιλούμε για το θεσμικό δεδομένου ότι εδώ θα κάνουμε συγκεκριμένε προτάσεις τρόπο με το οποίο θα προχωρήσουμε στο μέλλον και μεταξύ γυναικών, διότι εσείς, η Επίτροπος και εγώ, είμαστε γυναίκες και τρεις, δεν θα κάνω gentleman's agreement, γιατί είμαστε γυναίκε. gentlewoman's agreement. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια διαδικασία συνεργασία. Πάλι οι άντρε διαμαρτύρονται, όπω πάντα λέει η πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και πιστεύω ότι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον είναι κάτι το οποίο για τις εντολές διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες είναι κάτι το οποίο και θα πρέπει να συμφωνούμε μεταξύ μας δεδομένου ότι έχουμε την διαθεσμική συμφωνία και κυρίως διότι αυτό επιτάσσει πλέον και η συνθήκη της Λισαβόνας. Βεβαίως, οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να το συζητούμε μαζί σας για να είστε πάντα ενήμεροι και το ίδιο με την Επίτροπο, διότι όπως ξέρετε εμείς και με πραγματισμό, με πρακτικό πνεύμα και κυρίως με διαφάνεια θέλουμε να συζητούμε το οτιδήποτε. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και αυτό ακολουθούμε ως πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά ήθελα να πω και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με Τώρα θα συζητήσουμε το θέμα του κόκκινου τόνου και με την ε, Επιτροπή Ελέγχου και με τον κύριο Αμιλάτ και κλεισμένων των θυρών. Και ελπίζουμε ότι αύριο όλα θα γίνουν σύμφωνα με τις οι επιθυμίες όλων μας και οι συμφωνίες θα γίνουν έχοντας κυρίως κατά νου, όχι μόνο στο πλοίο εμείς, αλλά κυρίως έχοντας κατά νου το μέλλον του κλάδου. Ευχαριστώ. Bueno, eh, vamos a seguir la reunión. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μα με το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, το σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κώστερ, Διευθυντή τη Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου τη Αλληλίας του Βίγκο, σχετικά με τα αποτελέσματα του κοινού σχεδίου ανάπτυξη αλληλείας του ερυθρού τόνου του 2010 καθώς και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας το 2010. Bueno, como vamos relativamente regular de tiempo... Eh, Έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. ¿Arqueto? ¿O κύριος Κώστερ, όπω ξέρετε, έρχεται εδώ κάθε χρόνο και μας διηγείτε τι γίνεται στο Βίγκο, τι θα κάνει τον επόμενο χρόνο, Ποιε είναι οι προτεραιότητε. Θα μας μιλήσει τώρα και για τον ερυθρό που είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Και όπως είπε και η Επιτροπή, αύριο θα εγκριθεί και η εντολή για τον ερυθρό Φαντάζομαι ότι έχετε δει την προσωρινή έκθεση που έχει ετοιμάσει η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου, καθώς και το θέμα των δραστηριοτήτων. Δίνω το λόγο στον κύριο Κώστερ και μετά αν θέλετε θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεως. Όπως πάντα σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στις Βρυξέλλες από την μακρινή περιοχή του Βίγκο. Και ελπίζουμε ότι θα μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς γίνεται. Κάποιοι από εμά έχουν ήδη διαβάσει τις ε, εκθέσεις που μας αποστέλλετε, οι οποίες είναι άκρως ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκλησή σας να σας παρουσιάσω την έκθεση που αφορά τις δραστηριότητες της ε, ε υπηρεσίες μας, στην συνεργασία με το και την Επιτροπή για τον ε, έλεγχο της αλληλείας του ερυθρού τόνου, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός της πολιτικής μας. Ε, Βεβαίω είναι εξίσου σημαντικό μετά να θέσουμε σε εφαρμογή την πολιτική αυτή την οποία έχουμε καθορίσει. Διότι αν δεν γίνει σωστή η εφαρμογή της πολιτικής, οι στόχοι της πολιτικής δεν μπορούν να επιτευχθούν. Η κοινοτική μας υπηρεσία συνεργάστηκε με την Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να συντονίσει τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ε, κρατών μελών για τον αλληλεία του ερυθρού τόνου. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη νομική βάση που είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ερυθρού τόνου. Έχουμε την απόφαση της Επιτροπής που θεσπίζει ειδικό πρόγραμμα εποπτείας και ελέγχου Έχουμε την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρει ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι διαδικασίες, οι συγκριτικές αναλύσεις και ξέρουμε ότι σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη κάνουμε την ανάπτυξη του προγρήματος το οποίο θα θέσουμε σε παραγωγή βάσει αυτής της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τελικά έχουμε τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει τα το σχετικό πρόγραμμα αλίευσης του ερυθρού Η στόχη μας είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε συντονισμένοι μεταξύ μας τον κοινό έλεγχο και την, ε, να αναλάβουμε κοινές υπηρεσίες επιθεώρησης να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ο στόχος τελικά είναι ο έλεγχος, η εποπτεία και η επιθεώρηση στην θάλασσα, ε, στην ΙΚΑΤ, να έχουμε υποστηριστικές ε, εργασίες για την ε, ε, να ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, αλληλείας και ε, την όλη ε, παρακολούθηση της παραγωγής αυτής της διαδικασίας. Η κοινή μας στρατηγική είναι να μπορέσουμε να ασκήσουμε αυτό τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη θάλασσα την οποία έχουμε χωρίσει σε περιοχές και έχουμε για την επιθεώρηση ε, θαλασσίως τα κατάλληλα αεροσκάφη για να κάνουμε τις επιθεωρήσεις των ε, δραστηριοτήτων αλίας. Έχουμε πλοία τα οποία επίσης κάνουν τέτοιου είδους ε, εποπτεία και ε, έχουμε και επίγειους τρόπους επιθεώρησης. Η Επιτροπή συντονίζεται με την ε, κράτη-μέλη και με την κοινοτική μας υπηρεσία στα πλαίσια μιας μόνιμης ομάδας στην οποία εκπροσωπούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια αυτής της μόνιμης ομάδας ε, κάνουμε το σχέδιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, το σχέδιο δράσης. και τη διάρκεια του χρονιάς ε, παρουσιάζουν στα πλαίσια των συνεδριάσεων μας τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων των εποπτιών μας, συζητώνται τα αποτελεσματικά μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Έχουμε μία κοινή ε, ομάδα τεχνικής ε, ανάπτυξης και υποστήριξης. Έχουμε στα πλαίσια αυτής της ομάδας εθνικούς συντονιστές που ορίζουν τα κράτη-μέλη. Έχουμε συντονιστές από την ΖΕΦΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ομάδα. Έχουμε, έχουμε έναν, ε, κάθε φορά έναν εθνικό συντονιστή, ο οποίος συνεργάζεται με τους συντονιστές της EFCA, επιτόπου καθημερινά συζητούν βάση των πληροφοριών που λαμβάνομαι και των ε, αναφορών από τις επιθεωρήσεις επιτόπου όλα αυτά τα θέματα. Βάσει λοιπόν όλων αυτών των πληροφοριών αναλύουμε την κατάσταση για να είμαστε πάντα σίγουροι ότι τα σκάφη και τα αεροσκάφη επιθεώρησης ε, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του μπορούν να δουν τι ακριβώς γίνεται εκτός νομίμων πλαισίων για να αντιδράσουμε. Εδώ έχουμε την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το χρον... τη γραφική παράσταση την οποία βλέπετε. Έχουμε πληροφορίες όπως βλέπετε τα κράτη-μέλη για τις άδειες ε, αλίευσης. Έχουμε στοιχεία τεχνικά που φτάνουν την τεχνική ομάδα. Αναλύουμε τα δεδομένα που φτάνουμε για να μπορέσουμε να, να συντονίσουμε τις δράσεις και τις δραστηριότητε των ε, σκαφών επιθεώρησης και των μεθόδων που ακολουθούμε και Προσπαθούμε να συντονιστούμε όποια και να είναι η σημαία των αλληλευτικών στόλων και να ανοιχνεύσουμε οτιδήποτε παράνομο μπορεί να υποπέσει στην αντίληψή μας. Έχουμε προτεραιότητες ελέγχου 2010. Βλέπετε εδώ στο διαφάνεια αυτή πώς είχε η κατάσταση πριν από τις 15 Μαΐου, βασικά στην περιοχή της Μεσογείου όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες ε, ε, με παραγάδι για την αλλιεύση του ερυθρού τόνου. Βλέπετε τι γίνεται επίσης, τι ακριβώς γίνεται στο ψάρεμα με παραγάδι επίσης στην βόρεια πλευρά της Ευρώπης, στον, της Ευρώπης, στον Ατλαντικό, στη Βόρεια. όλα αυτά αφορούν, επαναλαμβάνω, τον ερυθρό τόνο. βεβαίως μιλούμε για παρασυρώμενα παραγάδια. Επίσης, βλέπετε τι ακριβώς συνέβη από 15 Μαΐου με τέλος Ιουνίου. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση επίσης από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο. Φέτος ήταν πολύ σημαντικό έτος για την αλληλεία του ερυθρού τόνου. Ένα μεγάλο ποσοστό των αλλιευμάτων αλλιεύονται σε αυτή τη μικρή περίοδο, 15 Μαΐου τέλος Ιουνίου. Επίσης προβλέπουμε κατάρτιση, κατάρτιση περιφερειακά στο Βίγκο. Εκεί που είναι η κοινοτική μας υπηρεσία έχουμε εθνικούς ε, εκπαιδευτές, υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Έχουμε οργανώσει εννέα εθνικές συνόδους κατάρτισης για την αλία του ερυθρού Έχουμε συζητήσει τα πλαίσια της κατάρτισης όλα τα σημαντικά θέματα. Οργανώσαμε επίσης ένα μάθημα για επιθεωρητές από άλλα συμβαλόμενα μέρη της ICAP. Οργανώσαμε επίσης ένα μάθημα στη Λιβύη για αξιωματούχους της χώρας αυτής και οι τελευταίες δραστηριότητες αναλήφθηκαν αιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις οργανώσαμε σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Ποιες είναι οι δραστηριότητες το 2010? Ε, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εστιάσεις πολλά αλλιευτικά σκάφη ακόμη. Τα... Είχαμε ε, φέτος σε σχέση με πέρσι πολύ λιγότερα αλλιευτικά σκάφη τα οποία αλλιεύουν. contracting parties, which was also a large έχετε εδώ ανα είδο τα αλλιευτικά σκάφη. Bold means. Dus we have been quite satisfied about the deployment of the pooled means. Dus we did not fully reach this what we. Δεν είναι πάντα τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις προβλέψεις. Επίσης πρέπει να πω ότι και οι κλιματικές ε, συνθήκες μας ε, επηρεάζουν. Πολλές φορές κάνουμε οικονομίες γιατί έχει κακό καιρό και δεν μπορούμε να στείλουμε τα λευτικά μας σκάφη και τα αεροσκάφη για επιθεωρήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν χωρίς να χάσουμε ε, την αποδοτικότητά μας πολλές φορές να κάνουμε και οικονομίες. όλες οι δραστηριότητες επιθεώρησης γίνονται σύμφωνα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν αλία μας. Για πρώτη φορά, επίσης, πρέπει να σας πω ότι εκ μέρους των κρατών μελών νοικιάσαμε και ένα ειδικό σκάφος επιθεώρησης, το Ζων και το σκάφος αυτό για 40 ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έκανε επιθεωρή στη Μεσόγειο κατά τη ε, διάρκεια της αλληλευτικής περίοδου. Με επιθεωρητές λοιπόν προσπαθήξαμε να κάνουμε τις σχετικές επιθεωρήσεις με την παρουσία συντονιστών και εκ μέρους της δικής μας υπηρεσίας. Βέβαια δεν μπορούν να κάνουν ε, τις επιθεωρήσεις όπως κάνουν οι ΆΕΚΑΤ για τους ζευγαρωτούς γρήπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το σκάφος μας ε, βοήθησε να κάνει πολλές επιθεωρήσεις στην περιοχή της Μεσογείου το καλοκαίρι. Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν τις δαπάνες. Η όλη διαδικασία ε, δεν ήταν εύκολη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να πληρώσουν για να ε, αναλάβουν αυτή τη δραστηριότητα και δεν είναι εύκολο να δίδει κανείς χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορέσαμε να οργανώσουμε το σκάφος αυτό για την επιθεώρηση. Πολλές φορές όμως είχαμε προβλήματα χρημάτων, διότι δεν έστειλαν εγκαίρως τη συμμετοχή του στο κρατημέλη και όπως καταλαβαίνετε ο πλειοκτήτης Μα πίεζε, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι προσπάθειε που κατέβαλαν για να χρηματοδοτηθεί αυτή η δραστηριότητα. Και ίσως στο μέλλον θα μπορούσε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και με χρηματοδότηση κοινοτική στα πλαίσια του σχετικού κανονισμού ο οποίος εγκρίθηκε το 2009. Then uh, Τέλος, να αναφερθούμε σε κάποιες από τις δραστηριότητές μας. Βλέπετε εδώ πέρα αρκετές. Καταρχάς, έχουμε τους επιθεωρητές, οι οποίοι βρίσκονταν στο σκάφος αυτό της επιτήρησης. Επιτηρήσεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, θα έλεγα. Το σκάφος αυτό βρίσκεται υπό τη διοίκηση της κοινή ομάδας επιθεώρησης που εργάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας μας. Η επιτήρηση, όπως ξέρετε, αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών και η τεχνική κοινή ομάδα εφαρμογής είναι ουσιαστικά απαρτίζεται από τους εθνικούς συντονιστές οι οποίοι κατευθύνουν το σκάφος αυτό στις διάφορες περιοχές όπου πρέπει να γίνουν ε, επιθεωρήσεις ή όπου θεωρείται ότι οι επιτηρήσεις θα είναι οι πιο αποτελεσματικές. Υπήρξε ένα μεγάλος βαθμός ευελιξίας για την ε, ανάπτυξη του, της ομάδας αυτής και είχαμε επιθεωρητές και συντονιστές από πολλά κράτη-μέλη. Επίσης, το σκάφος, αυτός μπορεί, το σκάφος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα κατάρτισης και κατά τη διάρκεια ενός ε, Σαββατοκύριακου ε, στο σκάφος αυτό ήρθαν και κάποιοι δημοσιογράφοι προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε και στον τύπο μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι κάνουμε και ιδιαίτερα για τον τομέα της αλίας του ερυθρού τόνου. Είδανε λοιπόν όλες τις δραστηριότητές μας και πώς εμείς παρεμβαίνουμε στην όλη διαδικασία της αλίευσης. Οι δημοσιογράφοι κατάφεραν λοιπόν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια όλου του Σαββατοκύριακου. Επίσης μπορείτε να δείτε εδώ πέρα τις επιθεωρήσεις που γίνανε στη θάλασσα, στην ξηρά. Φτάνουμε σε ένα σύνολο 630 επιθεωρήσεων. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει, όπως βλέπετε, το σύνολο των διαθέσιμων σκαφών που μας έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Από τα σκάφη αυτά, ένα μεγάλο μέρος συμμετείχε και σε επιθεωρήσεις που γίνανε το 2009 και όπως καταλαβαίνετε μέσω των επιθεωρήσεων εντοπίζουμε κάποιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Αυτές μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια αυτή. 34 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για κοινοτικά σκάφη και 18 περιπτώσεις για άλλα συμβαλόμενα μέρη στην ICAT. Σύνολο 52 λοιπόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Τα κοινοτικά αυτά σκάφη μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζουν γενικότερα μια καλύτερη συμμόρφωση σε σχέση με τα σκάφη από τρίτες χώρες. Κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα τώρα. Με τη συνεργασία των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουμε μια ανάλυση κινδύνου προκειμένου να επεξεργαστούμε όλη την εκστρατεία επιθεώρησης και προκειμένου να θέσουμε κάποιους στόχους κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και για να συμφωνήσουμε για το πώς θα διεξαγόταν η ε, όλη εκστρατεία. Τα κράτη-μέλη συνέβαλαν πολύ σημαντικά στο να συγκεντρώσουν πόρους, κατέβαλαν πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τις δραστηριότητες στις οποίες συμφωνήσαμε από κοινού στο κοινό σχέδιο εφαρμογής. Οι δραστηριότητες ελέγχου και επιθεώρησης διεξήχθησαν με την βοήθεια των ε, εθνικών συντονιστών, οι οποίοι συμμετέχουν στην ε, κοινή ομάδα τεχνικής εφαρμογής. Η συμβολή τους λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αν υπολογίσουμε τώρα κάποιους ε, δείκτες, δηλαδή τις περιπτώσεις εκείνες μη συμμόρφωσης σε σχέση με το σύνολο των επιθεωρήσεων, βλέπουμε ότι ο λόγος αυτός παρουσιάζει μία μείωση κατά 6%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλο και περισσότερα σκάφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον παρουσιάζουν ένα ποσοστό συμμόρφωσης σε σχέση με την κοινωτική νομοθεσία. Όπως σας είπα, το ποσοστό μη συμμόρφωσης έχει σημαντικά μειωθεί. Αν ε, καταλήξουμε λοιπόν σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την εκστρατεία του 2010, μάλλον παραθετικά να σας πω ότι το 2008 η υπηρεσία θεώρησε ότι ο λευτικός τομέας δεν θεωρούσε ως προτεραιότητά του την συμμόρφωση με τους κανόνες. Τώρα για το 2010 μπορούμε να πούμε ότι η συμμόρφωση έχει πλέον αυξηθεί τόσο από τα κοινοτικά σκάφη όσο και από τα σκάφη τρίτων χωρών. Καταβάλλονται δηλαδή από όλου όλο και περισσότερε προσπάθειε προκειμένου να τηρήσουν τι απαιτήσει, προκειμένου να δείξουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό συμμόρφωση. Επίσης, είδαμε ότι υπήρχαν πολλά σκάφη τα οποία μετά την ολοκλήρωση της αλληλευτική προσπάθειας, ακόμα και όταν δεν είχαν φτάσει το ανώτο ποσοστό προβλέπεται από την ποσόστοση, αποφάσισαν θελοντικά να επιστρέψουν στους λιμένες και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα παραπάνω δείγμα βούλησης για συμμόρφωση. Επίσης, ε, παρατηρήσαμε κάποιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά τα τάξ. Στις ε, περισσότερες ε, περιπτώσεις είδαμε ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη καταγραφή της ελευτικής προσπάθειας στο μητρό του σκάφους. Και στον τομέα αυτό είδαμε ότι υπάρχει μία βελτίωση, ωστόσο πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό συμμόρφωσης και σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Eh, ευχαριστώ πολύ. Πριν να περάσουμε στη συζήτηση, θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων σας και τον υπόλοιπο χρόνο τον αφιερώσουμε στη συζήτηση. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων είναι το 2011. Να μας το εξηγήσετε και μετά θα αρχίσουμε τη συζήτηση και ο καθένας θα σας κάνει την ερώτηση που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Madam Chairman. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμα εργασίας της υπηρεσίας μας, του οργανισμού, για το 2011 και την περίοδο 2011-2015 Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον έλεγχο που εγκρίθηκε το 2009, ο οργανισμός θα πρέπει δηλαδή να καταρτίζει πολιετές πρόγραμμα εργασίας για πέντε χρόνια. Αυτό προβλέπεται και είναι ένα κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας δηλαδή. Κάθε φορά έχουμε το επόμενο πολιετές και τις ε, πενταετής ε, προοπτικές και τον απολογισμό δραστηριοτήτων επίσης. Τώρα, για το, την επόμενη πενταετία, το πρόγραμμα εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή του Οργανισμού και κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, την Κομισιόν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται οι προτεραιότητες του οργανισμού για την επόμενη περίοδο. Οι προτεραιότητες βέβαια πρωτίστως είναι ότι πρέπει να ε, συμβάλλουμε στις δραστηριότητες IUU, δηλαδή να καταπολεμήσουμε την παράνομη άναρχη λαθρέα αλληλεία όπου και συμμετέχει ο οργανισμός ε, μαζί με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη σε, αυτό, το, σε αυτές δραστηριότητες για να σταματήσουν οι παράνομες εισαγωγές. Ο κανονισμός ε, ισχύει από την αρχή αυτού του έτους. Ο οργανισμός ε, κάνει κατάρτιση των εθνικών επιθεωρητών και βοηθάει επίσης την Κομισιόν με ελέγχους σε τρίτες χώρες για να διαπιστωθεί αν το σύστημα πιστοποίησης κάτσε σε τρίτες χώρες τηρείται. Λίγος πολύ σωστά. Και εκεί ο οργανισμός μας μαζί με την Κομισιόν κάνει ελέγχους και στα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται δηλαδή αυτό, για να διαπιστωθεί η κατάσταση και όπως σας είπα και στις τρίτες χώρες ε, για το σύστημα GATS. Μετά στον επιχειρησιακό συντονισμό θα, δραστη, θα δραστηριοποιούμε θα στους ίδιους τομείς όπως και τώρα Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Μεσόγειο και νάφο ναύτα αέρια, ε, περιοχή και Ατλαντικό δηλαδή και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων θα αναβλώσουμε και ένα ε, σκάφος επιθεώρησης, αν υπάρχει δυνατότητα οικονομική. Τώρα, εκτός από τις δραστηριότητες επιχειρησιακού συντονισμού, ε, έχουμε τη δημιουργία ικανοτήτων ως προτεραιότητα που βοηθάει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν και να υλοποιούν την κοινή αλλιευτική πολιτική με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο. Ένας τομέας όπου θα αναπτύξουμε εκπαίδευση είναι στους εθνικούς επιθεωρητές για να διασφαλίσουμε ότι οι επιθεωρητές στην Αλία από όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν καταρτιστεί σωστά για να ξέρουν πώς θα εφαρμόζουν την κοινή αλληλευτική πολιτική με τρόπο ενιαίο, να είναι εκπαιδευμένοι με τον ίδιο τρόπο. Θα έχουμε δηλαδή ένα βασικό αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτό ε, έχει αρχίσει και θα το αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια περισσότερο. Επίσης αν το ζητήσουν τα κράτη-μέλη θα παράσχουμε επικούρηση στην εθνική εκπαίδευση. Αλλά η βασική δραστηριότητα θα είναι να καταρτήσουμε το βασικό αναλυτικό πρόγραμμα και να οργανώσουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εθνικούς επιθεωρητές και τους εκπαιδευτές. Επίσης, ε, χρειάζονται δεδομένα ενημέρωση για τα δεδομένα, ενημέρωση για την ε, αλληλεία πριν από λίγα χρόνια το ελεκτικό συνέδριο υπέβαλε μια έκθεση που δεν ήταν και τόσο θετική σε σχέση με το πώς διατίθενται τα δεδομένα ε, για τη λήψη αποφάσεων. Ο νέος κανονισμός για τον έλεγχο ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και τα σχετικά προβλήματα. Ο νέος κανονισμός όμως για τον έλεγχο θα πρέπει να εφαρμόζεται. Και εμείς συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ώστε να φροντίσουμε να δούμε πού πρέπει να βελτιώσουν τα κράτη-μέλη, τα εθνικά συστήματα δεδομένων, τις βάσεις δεδομένων και να φροντίσουμε να γίνουν οι επενδύσεις για τη βελτίωση των βάσεων δεδομένων που πρέπει να γίνουν για να είναι και διαλειτουργικό το σύστημα και πιο εναρμονισμένο ώστε να ε, διευκολύνεται η ανταλλαγή των ε, δεδομένων και να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για κοινά σχέδια, προγράμματα ανάπτυξης ε, και να έχουμε αυξημένη αποτελεσματικότητα. Αυτό θα πάρει κανένα δύο χρόνια. Θα είναι πολύ δραστήρια δηλαδή μαζί με την Κομισιόν στα δύο αυτά επόμενα χρόνια σε αυτό το τομέα μαζί με την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τι εξηγήσει κύριε Κώστερ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριο Ρωμέρο πρώτος. Ευχαριστώ, και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Κώστερ που ήρθατε και μας εξηγήσετε όχι μόνο το πρόγραμμα αλλά και τα αποτελέσματα των κοινών δράσεων για τον έλεγχο του ερυθρού τόνου μέχρι τώρα. Τρία βασικά σχόλια ή ερωτήσεις από μένα. Πρώτον, μετά τις τελευταίες πληροφορίες που έδωσε η ίδια η ICAT, βλέπουμε, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, ότι το σύστημα της ανιχνευσιμότητας ή ιχνηλασιμότητας ε, και όχι μόνο ο έλεγχος αλλά και η υποβολή δεδομένων ε, αναλαμβάνεται από τα κράτη-μέλη, τα συμβαλόμενα μέρη. Για να το πούμε ήπια, το σύστημα είναι δυσλειτουργικό. Ε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε όχι μόνο την ε, ικανότητα ελέγχου και δυναμικό ελέγχου, αλλά να δούμε και την ωφελημότητα του συστήματος του ίδιου, όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα. Τώρα, αν δούμε διάφορες εκθέσεις που υπέβαλαν οι επιθυρητές, αλλά και τις επίσημες εκθέσεις που δίνει ο ίδιος ο κλάδος, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αναντιστοιχίες που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά για την ορθότητα του ίδιου του συστήματος. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Είδαμε τις συγκεκριμένες βελτιωτικές προσπάθειες του οργανισμού για τον έλεγχο μέρους του συστήματος. Αλλά θα πρέπει να καλυφθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ο έλεγχος κάποιων συμβαλωμένων μερών της ε, ICAT θα ε, συγκρίνεται ευνοϊκά και με τη δραστηριότητα άλλων συμβαλωμένων μερών. Είπατε ότι μειώθηκαν οι διαφορές. Αυτό βέβαια καλό πράγμα είναι, αλλά μπορείτε να εξειδικεύσετε. Δεύτερον, επίσης που συγκεκριμένο, μιλήσατε για το ρόλο του σκάφους αυτού του Ζαν Σαρκό. Φαντάζομαι ότι ένα σκάφος για ολόκληρη τη Μεσόγειο δεν φτάνει, δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα με αυτό. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος για το πώς αντιδράτε, ας πούμε, αν υπάρξει κάποια υποψία. Ποια είναι η ικανότητά σας, η ικανότητα που υπάρχει να εντοπιστούν κάποιες παράνομες ή νόμιμες δραστηριότητες στη θάλασσα. Ποια είναι η, ποιο είναι το δυναμικό ελέγχου του σκάφους, πώς μπορεί να ελέγχει δηλαδή τις θαλάσσιες δραστηριότητες, για να έχουμε κι εμείς μια ιδέα πόσο αξιόπιστα είναι τα ε, δεδομένα που ε, παρέχει το σκάφος. Τρίτον και τελευταίο. Είναι κάποιοι περίεργοι και δυσανάγνωστοι πίνακες εις ό,τι αφορά την ε, μη συμμόρφωση. Σε σχέση με την επόμενη ΆΙΚΑΤΑ στο Παρίσι. Αν συζητήσουμε τα τάκ που θα πρέπει να εφαρμοστούν, να ισχύσουν, θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέχρι τώρα η εφαρμογή των κανόνων που έχουν συμφωνηθεί και που χρειάζονται δεν έχουν εφαρμοστεί απόλυτα. Ας μιλήσουμε για τη μαύρη αγορά, ας πούμε, να αν είναι μεγαλύτερη αυτή τελικά από ό,τι νομίζαμε, ο υπολογισμός των τάξ στο Παρίσι, αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη. Πολύ συγκεκριμένα ρωτώ λοιπόν, πώς φαντάζεστε την αξιολόγηση ή την πιστοποίηση του συστήματος. Αν δηλαδή είναι καλό αυτό και μπορούμε να μιλάμε για καινούρια τάκ και για τους 13.500 τόνους ή θα πρέπει να περάσουμε σε πιο δραστικά μέτρα και αποφάσεις κάποιο μορατόριουμ ή μηδενικό τάκ για κάποιο διάστημα. Ο κύριος Ρήμες. Κυρία Ρήμες, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή. Έχουμε νούμερα, έχουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε τώρα για την αρχή ελέγχου CFSA και το πρόγραμμα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Με ενδιαφέρει όμως να μου πείτε τι πιστεύετε για τον, την επιτυχία αυτών των μέτρων. Πόσο επιτυχής ήταν η εφαρμογή του σχεδίου σε σχέση με το στόχο του καλύτερου ελέγχου των αλληλευτικών δραστηριοτήτων για τον τόνο. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις και ή είχατε προβλήματα κατά την εφαρμογή του σχεδίου σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαβίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Κώστερ. Γνωρίζετε φαντάζομαι τις νέες αυτές ιστορίες που δημοσιεύονται ε, στα ΜΜΕ και στις εφημερίδες σε όλη την Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, από μεγάλες εφημερίδες τα ψάξαν τα θέματα οι δημοσιογράφοι και λένε ότι όταν μιλάμε για τα αποθέματα ερυθρού τόνου και τις προσπάθειες για αυτά υπάρχει ελλειπή ενημέρωση. Και τέλος πάντων τα μέτρα δεν πραγματοποιήθηκαν όπως έπρεπε. 80% αυτών ε, των θυναλιευτικών δεν λειτουργούν σωστά, δεν έχουν πληροφορίες για τα εισαγόμενα είδη, λείπουν, λείπουν πολλές ε, σημαντικές πληροφορίες και απαραίτητες. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό πράγμα. Και θα ήθελα τα σχόλιά σας σχετικά με αυτές τις καινούργιες ε, ε, ιστορίες που, που γράφουν τα ΜΜΕ. Βέβαια και από τα λεγόμενά σας επιβεβαιώνονται κάποιες γιατί η πιο σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης αφορά τα σωστά μητρώα, την ε, τήρηση ε, ε σε σχέση με τα αλλιεύματα. Ε, θέλω επίσης να ακούσω και πάνω σε αυτό την ανάλυση τη δική σας. Πώς γίνεται να λείπουν ή να είναι ελλειπή τα στοιχεία. Ποιος φταίει, τα κράτη-μέλη, τα συμβαλόμενα μέρη που δεν παίρνουν στην αποστολή τους τα σοβαρά για να φροντίσουν ότι όλοι και οι επιχειρήσεις και οι αλληλείς θα πρέπει να κάνουν ό,τι πρέπει για να συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα με σωστό τρόπο. Πείτε μας λοιπόν τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κώστερ. Α, χαρήκαμε πολύ πρέπει να πω την επίσκεψή μας στο Βίγκο και χαρήκαμε που είδαμε ότι υπάρχει τέτοια προσοχή από το προσωπικό σας στο ζήτημα του ερυθρού τόνου. Συνεχίζοντας όμως σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λοβίν, Χθε στους Sunday Times γινόταν μία έρευνα, γινόταν μία αναφορά σε μία έρευνα της WWF όπου λέγεται ότι υπάρχουν ε, πολλά σκάφη τα οποία δεν συμπληρώνουν σωστά τα έγγραφα αλλιευμάτων όσον αφορά τον ερυθρό τόνο, ότι υπάρχουν ε, γενικά πολλές ε, παρατυπίες και θα έλεγα ακόμα και εγκληματικές δραστηριότητες όσον αφορά την αλία. Και όλα αυτά πιστεύω ότι έρχονται σε αντίθεση με αυτά τα οποία εσείς μας παρουσιάσατε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη για αυτά τα σχόλια του τύπου. Επίσης, ενδεχομένως να με είχατε ακούσει να λέω νωρίτερα, όταν παρούσε εδώ ήταν η κυρία Evans, ότι έχω κάποιες ανησυχίες ε, όσον αφορά το σκουμπρί. Ξέρω ότι ε, εσείς ε, ασχολείστε πολύ περισσότερο με τον ερυθρό τόνο και με τον περιορισμένο, τους περιορισμένους σπόρους γι' αυτό. Η ISIS πάντως λέει ότι η Ισπανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει ένα 286% των μικροποσοστώσεών τους και νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να τα είχατε καταγράψει κάπως στο Βίγκο. Μόλις ότι ασχολείστε με τον τόνο, νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να ασχοληθείτε κάπως και με το σκουμπρί. Ξέρω τουλάχιστον ότι στη Σκωτία το 2004 ε, υπήρχαν σκάφη, πλειοκτήτες ε, που ε, έλαβαν τεράστια πρόστιμα για την παράτυπη δραστηριότητά τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει η αλίευση οποιοδήποτε ψαριού να καταγράφεται Είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό λοιπόν ότι στη δική μου εκλογική περιφέρεια κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ενδεχομένω να συμβαίνουν παράνομε εκφορτώσει και σε άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικό είναι η παράνομη αυτή δραστηριότητα να καταγράφεται. Θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλιά σα. Διαβάζω τον κατάλογο και θα την κλείσω, διότι μετά έχουμε και άλλα θέματα στη μερίσια διαδοχή. Κύριε Άντοψ, Κάντεξ, Αντρέ Βαρέα, Αρσένη, Αντόκ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι πρέπει να έχουμε και την συνεδρία σκυκλισμένα των θυρών και μετά έχουμε και τη συνάντηση των συντονιστών. Κύριος Καντέκ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Κόσνερ για την παρουσίασή σας. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα μιλήσατε για 34 παραβάσεις που διαπιστώσατε. Τι είδους, Γιατί τι είδους παραβάσεις μιλάτε. Οι ίδιες ήταν διαφορετικές Περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Επίση, όπως είπε και ο κύριος Στίβενσον, και εγώ αντιδρώ μετά από αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος Ισαμπέλα όσον αφορά τα αποκόμματα τύπου τα οποία διαβάσαμε. Και είπε ότι πρόκειται για ε, άρθρα που έγιναν ε, μετά από έρευνα και άρθρα τα οποία έγιναν ε, στα πλαίσια μη κυβερνητική οργάνωσης. Διαρωτώ με δεδομένου ότι όχι στον τομέα τη αλλά και σε πολλούς άλλους τομεί. έχουμε εκπροσώπους τύπου που κάνουν έρευνες όλο και περισσότερο σε πολλούς τομείς. Τώρα έχουμε να κάνουμε με την αλληλεγγύη συγκεκριμένα και έχουμε στο Βίγκο μία κοινοτική υπηρεσία ελέγχου. Εγώ μάλλον έχω πρέπει να προσέξω τι μου λέτε εσείς, που φαντάζομαι ότι είστε σοβαροί και επαγγελματίες και κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Δεν θέτω σε αμφιτητήσει βεβαίως την δουλειά που κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κυρίως η WWF, αλλά με ανησυχεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, κάθε φορά στον τύπο δημοσιεύονται διάφορα άρθρα και σχόλια, όχι μόνο στην Αλία, αλλά και σε άλλους τομείς, χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικές συγκεκριμένε πληροφορίες και ενημέρωση. Είδαμε πολλές φορές ε, και διάφορα ντοκιμοντέρ και στην τηλεόραση. Δεν το βλέπουμε μόνο στο γραπτό τύπο. Στην τηλεόραση πολλές φορές ή στο ραδιόφωνο κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες θα ήθελα να μου πείτε εσά ποια είναι η άποψή σα. Φαντάζομαι ότι ξέρω τι έχετε να πείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα ήθελα να ε, υπογραμμίσω ότι εμείς εμπιστευόμεθα την κοινοτική υπηρεσία λαχπιότητας διαφορετικά. Τι, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλέον κανένα. Τι κάνουμε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Είπατε ότι ένα μεγάλο μέρος της εργασίας σας αφιερώνεται στην ε, εκπαίδευση για να υπάρχουν ενιαία κριτήρια. Σωστό είναι αυτό. Είπαν κάποιες συνάλληψεις ερωτήσεις ότι πολλές φορές ε, βασίζεστε στην καχυποψία που υπάρχει ίσως πολλές φορές ε, και στις υποψίες που υπάρχουν μεταξύ όλων. Και πολλές φορές υπάρχουν και τα δημοσιεύματα στον τύπο από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι ερωτήσει μου είναι πώς επιπαληθεύονται τα δεδομένα και πόση διαφάνεια, πόσο στα πλαίσια της διαφάνειας μπορούμε να έχουμε ε, εμπιστοσύνη στα δεδομένα που κυκλοφορούν ώστε να μην πέσουμε στις παγίδες των διαφόρων άρθρων. Δεύτερον, Δεδομένου ότι εσείς είπατε ότι ε, στην επόμενη περίοδο από τα κριτήρια τα οποία ε, θα ακολουθήσετε είναι το θέμα της κατάρτισης. Ποιες είναι οι χώρες που θέλουν να έχουν ενοποιημένα, δηλαδή κοινά κριτήρια και θέλουν επίσης να ε, συμμετάσχουν στην κατάρτιση. Ο κύριος Αρσένης. Ε, Κύριε Κώστερ, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Θα ήθελα και εγώ να ακούσω τις, ε, τα δικά σας σχόλια για τα άρθρα αυτά, τα οποία φαίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικά για όλους μας. Επίσης, αναφερθήκατε, και το είπε αυτό και ο κύριος Καντέκ και συμφωνώ μαζί του, σε διάφορες ε, παραβάσεις. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω ποιες παραβάσεις δεν καταφέρατε να εντοπίσετε, αλλά ακόμα και στις 18 αυτές κοινοτικές περιπτώσεις θα λέγαμε στις 18 αυτές μη συμμορφώσεις, ποιες περιπτώσεις είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι σαφώς θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό επίπεδο συμμόρφωσης για τις αποφάσεις της ICAT. Πρόκειται να γίνουν κοινή έλεγχη και με άλλα κράτη της Μεσογείου. Και σκέφτεστε να αυξήσετε την διαθεσιμότητα πόρων προκειμένου να διεξάγονται τέτοιοι έλεγχοι. Γιατί νομίζω ότι ε, οι έλεγχοι τόσο για κοινοτικά σκάφη όσο και για σκάφη κρατών της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στοχεύουν στο να έχουμε τελικά μία βιώσιμη αλία και βιώσιμα αποθέματα. Ευχαριστώ. Στην Έκθεση τη ε, κοινοτικής υπάρχει ένα πίνακα στον οποίο βλέπουμε αναχώρα ποιο έκανε παράβαση, τι είδου, τι γίνεται. Υπάρχει ένας ε, πολύ καλός ε, επεξηγηματικός ε, πίνακας. Κυρία Χάντου, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις μετά από αυτά τα οποία ερώτησε ο κύριος Στίβενσον. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνει για να επιθεωρήσει τουλάχιστον εφέτος τις δραστηριότητες αλληλείας ε, των ε, η δική σας κοινοτική υπηρεσία. Επίσης μπορείτε να μας πείτε εάν έχετε σχέδια συμμετοχής ε, ε, ελέγχου που θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει ε, με την αλληλεία της Ισλανδίας και τις ποσότητες των αλλιευμάτων μακροπρόθεσμα. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει σχετική συμφωνία και ότι όλα είναι πολύ αμφιλεγόμενα. Κύριε Κώστερ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έγιναν. Thank you very much, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, στο ερώτηση του κυρίου Ρέμοβα, την ιχνηλασιμότητα, τα BCDs όπως λέγονται. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία αναφέρεται και στην ιστορία αυτού του δημοσιογράφου που το, δήμος το Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε και στο BBC και τις άλλες εφημερίδες. Η τεκμηρίωση της BCB είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντική για τον έλεγχο της αλίευσης ερυθρού υπήρχαν μεγάλα προβλήματα με τον ερυθροτόνο και κατά τη διάρκεια της ακρόασης που έκανε η Επιτροπή Ελίγειας το 2007. Όταν εσείς δηλαδή ε, καλέσατε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να γίνει μια ενημέρωση για τον ερυθρότονο. Υπήρχαν πολλά πράγματα που ήταν λαθασμένα από αυτό που γίνονταν. Διάρκεια αυτής της ακρόασης προσπαθήσαμε κάπως να διορθώσουμε την όλη κατάσταση και να κάνουμε ένα σύστημα εποπτείας πολύ καλό για να σώσουμε τον ρυθμό τόνο. Αρχίσαμε εμείς να συντονίζουμε τις δραστηριότητες των κρατών μελών το 2008. Συνεργαστήκαμε στενά με τα κράτη-μέλη και την Κομισιό από την ε, κοινωνική μας υπηρεσία για να κάνουμε καλύτερους ελέγχους από το 2008. Βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο σήμερα δηλαδή. Πολλοί ερώτησαν αν είναι επιτυχής δραστηριότητές μας. Στην... Φέτος θα με εξέπλησε πάρα πολύ εάν υπήρχε υπεραλίευση και αν είχαν ξεπεραστεί οι ποσοστώσεις. Κανένας δεν μπορεί να πει βέβαια ότι κάτι δεν είναι αδύνατο, αλλά πιστεύω ότι το 2010 έχει γίνει σωστή αλήθεια. Το 2007 σε αυτή την ακρόαση υπήρχε και βιολόγος από την ICAT που είπε ότι τα πραγματικά αλλιεύματα ήταν διπλάσια από τις ποσοστώσεις. Ήταν τότε 30.000 τόνοι. Νομίζω ότι έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη βελτίωση από τότε. Η ιστορία αυτή της VVF ε, και αυτό το οποίο είπαν οι δημοσιογράφοι στο BBC είναι ότι κοίταξαν όλα τα σχετικά έγγραφα που μπορούσαν να βρουν για τις αλληλευτικές δραστηριότητε του ερυθρού τόνου από το 2002, 2000, ε, από το 2008, 2009 και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν βασίστηκαν σε έγγραφα του 2010. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνεί με την εικόνα που παρουσίαζε και πες και πρόπερση εδώ στο Κοινοβούλιο, όταν σας είπα ανοιχτά εδώ ότι η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική. Και στην πρώτη έκθεση την οποία αποστήλαμε για τις δραστηριότητες του Ερυθρού Τόνου είπαμε ότι προφανώς δεν ήταν μία από τις προτεραιότητες του αλληλευτικού κλάδου να συμμορφωθεί με τους κανόνες. Από εκεί ξεκινήσαμε. Προχωρούμε και πάμε σε μια κατάσταση η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη. Δεν θα σας πω βεβαίως σήμερα ότι η κατάσταση το 2010 είναι απολύτως ικανοποιητική. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα και με τα έγγραφα και με τα BCDs, αλλά βεβαίως έγινε σαφής, υπάρχει σαφής βελτίωση και το 2008 είχαμε μια κατάσταση που βελτιώθηκε το 2009 και το 2010 είχαμε βελτιωμένη κατάσταση σχέση με το 2009, 10 σχέση με το 2009 και συνεχίζουμε. Στην παρουσίαση αυτή που έγινε στο BBC επέκριναν τα BCDs που είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τους ελέγχους. Εμείς Ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει πολύ καλή τεκμηρίωση για να μπορεί κανείς ε, το, να ελέγχει την, το σύνολο της επιτρεπόμενης ποσότητας αλλιεύματος. Έχουμε οργανώσει ε, επιθεωρήσεις, στο BCD και τα σχετικά βιβλία στα οποία εγγράφονται οι καταγράφονται οι αλλιευόμενες ποσότητες βρίσκονται στα αλλιευτικά σκάφη και τα πρέπει να παρακολουθεί κανείς την κατάσταση στα έγγραφα σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας. Πολλές φορές είχαμε λυπή ενημέρωση των σχετικών βιβλίων και για τα τάξ και για τις ποσοστώσεις. Το 2010 βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση Άρα νομίζω ότι υπάρχει, έχει γίνει προτεραιότητα τα σχετικά έγγραφα να ενημερώνονται σωστά. Επίσης, όταν επιθεωρούμε αλλιευτικά σκάφη άλλων κρατών της ΑΚΑΤ, βλέπουμε ότι έχουν γίνει επίσης για την συμπλήρωση των σχετικών βιβλίων και μητρών που καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες βελτιώσεις. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει η χνηλασιμότητα για τον αριθμό τόνων αρχίζει από τη στιγμή της αλίευσης μέχρι τη στιγμή που φτάνει στην Ιαπωνία, στο πιάτο του κάθε Ιαπωνέζου. Γιατί όπως ξέρετε το 89% του ερυθρού τόνου πηγαίνει στην Ιαπωνία και θα πρέπει να ελέγχουμε πλήρως την διαδικασία ιχνηλασιμότητας. Από την αρχή ως το τέλος. Στην έκθεση του BBC βλέπουμε ότι σταμάτησε τις εισαγωγές η Ιαπωνία, δεδομένου ότι υπήρχαν προβλήματα με το BCD, με τα σχετικά έγγραφα που αφορούσαν την αλίευση του ερυθρού Άρα είπαν οι Ιαπωνέζοι δεν θα εισάγουμε πλέον εάν υπάρχουν προβλήματα με το BCD, το Blue Fin Tuna Catch Document. Και βεβαίως θα πρέπει να ενεργούμε όλοι σωστά για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή τη δραστηριότητα. Τώρα, μου, μου ζητήσει κάποιο φοβεί για το Ζων Σαρκό, για το σκάφος αυτό επιθεώρησης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σκάφη επιθεώρηση από τα κράτη-μέλη που αφορούν την, επιθεώρηση για την αλίευση του ε, ερυθρού Προσθέσαμε το σκάφος αυτό ως κοινοτικό σκάφος επιθεώρησης, ώστε να είναι, αν θέλετε, και ένα ουδέτερο βήμα. Και υπάρχει και βεβαίως ε, η βούληση να έχουμε και συνεργασία με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναφέρω το παράδειγμα της Λιβύης, δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή διαδικασία. Ελπίζουμε του χρόνου θα μπορέσει να γίνει. Αλλά όπως σας είπα είναι κάτι το οποίο στοχεύει και στη συνεργασία με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την επιθεώρηση σωστά. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο και παραγωγικό το ότι είχαμε τον Ζων Σαρκό και επιθεωρητές από όλα τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν υπό την ε, αιγίδα αυτής της κοινή τεχνικής ομάδας, εργάστηκαν όλοι σωστά και βρήκανε και κάποιες παρατυπίες και εκείνοι. Στη συνέχεια, όσον αφορά την πολιτική μας, η ερώτησή σας ήταν ε, η... ο πίνακας αυτός για τις παραβάσεις. Υπάρχει ένας πίνακας στην έκθεση. Μπορείτε να δείτε τα σκάφη και από ποια χώρα προέρχονται, τα σκάφη αυτά τα οποία έχουν προχωρήσει σε παραβάσεις. Το καλύτερο θα ήταν να συμβουλευτείτε τον πίνακα αυτό για να καταφέρετε να δείτε όλες τις παραβάσεις και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να μιλήσω αυτή τη στιγμή για την πολιτική, αν θα πρέπει να μειωθεί το ΤΑΚ ή αν θα πρέπει να έχουμε ένα μορατόριουμ. Εμεί ουσιαστικά μέσω τη υπηρεσία μα προσπαθούμε να συντονίσουμε τι δραστηριότητε, επιθεώρησης και επιτήρηση των κρατών μελών. Επομένω δεν δύναμε να σχολιάσω το ζήτημα τη πολιτική που θα πρέπει να ακολουθεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο ερώτημά σα, πόσο επιτυχεί είμαστε Κοιτάξτε, υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση που βαίνει προς τη βελτίωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι τα πράγματα είναι τέλεια του 2010 και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σαφώς όμως υπάρχει μια θετική τάση, υπάρχουν συνεχείς ε, αποδείξεις ότι όντως προχωράμε προς ε, την ε, επιτυχία και υπάρχουν σαφές βελτιώσεις όσον αφορά το όλο πνεύμα της συμμόρφωσης όλο και περισσότερα λεπτικά σκάφη τείνουν να συμμορφώνονται. Σαφώς υπάρχει το ζήτημα των ζευγαρωτών γρήπων, αλλά και το πρόβλημα αυτό έχει παρουσιάσει μείωση. Τώρα, η ιστορία του BBC. Όπως σας είπα, δεν υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία στην ιστορία αυτή. Ήδη γνωρίζαμε το γεγονός αυτό. Το άρθρο του BBC βασίζεται σε πράγματα που έχουν συμβεί το 2008, 2009, αλλά και στο παρελθόν. Και οι πληροφορίες από την εκστρατεία του 2010 δεν περιλαμβάνονται μάλιστα στο άρθρο. Το άρθρο επίσης αυτό επιβεβαιώνει τις βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει, γιατί λέει ξεκάθαρα ότι ε, έχουν ε, επέλθει βελτιώσεις. Λέει επίση όμως και το άρθρο ότι υπάρχουν ακόμα πολλά κενά τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Επομένως, είναι συζητήσιμο αν θέλετε το πόσο χωλαίνει το σύστημά μας ή το πόσα νομικά κενά αυτή τη στιγμή παραμένουν. Αυτό μπορώ να πω εγώ και να επιβεβαιώσω είναι ότι ε, σαφώς συνεχώς βελτιωνόμαστε και η μελέτη καταδεικνύει ότι όντω υπάρχει αυτή η συνεχή βελτίωση. Ουσιαστικά μα ενθαρρύνει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο προκειμένου να καταφέρουμε να ελέγξουμε πλήρω όλο το τομέα τη αλεία. Όσον αφορά τώρα το σκουμπρί και την υπηρεσία μας που βρίσκεται στο Βίγκο, κοιτάξτε, Σίγουρα τα πράγματα εδώ πέρα είναι κάπως πιο δύσκολα. Ο κύριος Στίβενσον αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στην αλία για το σκουμπρί στον κόλπο της Γασκόνη, στα δυτικά λοιπόν ύδατα, καθώς επίσης και αναφέρθηκε στον αλλιευτικό αυτό στόλο, ο οποίος απαρτίζεται κυρίως από μικρά αλλιευτικά σκάφη. Πρόκειται λοιπόν για κάποια μικρά λευτικά σκάφη τα οποία αλλιεύουν σκουμπρί, κυρίως τράτης για παράδειγμα. Δεν υπάρχει στα δυτικά ύδατα κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο επιτήρησης για τη δική μας υπηρεσία. Ενδεχομένως θα έπρεπε εδώ πέρα να έχουμε ένα κοινό σχέδιο ανάπτυξης ομάδων επιτήρησης και ενδεχομένως θα ήταν θετικό να ενθαρρύνουμε τον ελευτικό κλάδο να αποδεχθεί ένα τέτοιο σχέδιο επιτήρησης και στην περιοχή αυτή, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε στην περιοχή αυτή ένα καλύτερο επίπεδο ελέγχου. Σαφώς το χρειαζόμαστε αυτό. Υπάρχουν αντικρώμενες καταστάσεις μεταξύ των διαφόρων ελευτικών στόλων, επομένως είναι πολύ καλό να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα επιτήρηση και εκεί. Όπω γνωρίζετε όμω, τα μέσα και οι πόροι τη υπηρεσία μα είναι περιορισμένα. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα κοινό σχέδιο επιχείρηση και στην περιοχή αυτή. Ουσιαστικά αυτό θα εξαρτηθεί από του πόρου που θα πρέπει να έχουμε προκειμένου να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σχέδιο και στην περιοχή. Σαφώ θα θέλαμε να ασχοληθούμε με την επιτήρηση και στα δυτικά ιδία, αλλά δεν έχουμε ακόμα του απαραίτητου πόρου για κάτι τέτοιο. Αυτά όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Στίβενσον. Λάβαμε και την επιστολή του και την επιστολή του κυρίου Τότ και κάποιων άλλων βουλευτών όσον αφορά το σκουμπρί πάντα. Από προσωπική μου λοιπόν περιέργεια είδα την επιστημονική έρευνα που έχει γίνει και ενημερώθηκα λίγο περισσότερο για το ζήτημα. Ε, διάβασα λοιπόν τις επιστημονικές έρευνες, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα πιο μπερδεμένος ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της αλίας ε, για το σκουμπρί στα ειδικά ύδατα. Έχουμε εδώ πέρα έναν στόλο, ο οποίο ε, αλλιεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρτίζεται, όπως σας είπα, από, κάποιες, από κάποια πολύ μικρά λευτικά σκάφη, τα οποία έχουν ε, ποσοστώσει σε καθημερινή βάση και η κατανάλωση είναι κυρίω και αυτή σε καθημερινή βάση. Έχουμε μια κατανάλωση νοπών ψαριών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε κάποια αριθμητικά δεδομένα τα οποία δεν αποκρίνονται απολύτω στην πραγματικότητα. Βέβαια, όταν είδα ότι μέσα σε ένα έτος διπλασιάστηκε η αλίευση, ενώ είχε μείνει σταθερή για πάρα πολλά χρόνια, και το να διαβάσω αυτή τη στιγμή στην επιστημονική έρευνα ότι ε, δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά ο λευτικός στόλος, ουσιαστικά δεν έχουν προσθεθεί περισσότερα σκάφη, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αυτά με μπερδεύουν ακόμα περισσότερο. Όπως σας είπα όμως, η υπηρεσία μας δεν έχει ένα κοινό σχέδιο επιχείρησης για την γεωγραφική αυτή περιοχή. Η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από λίγο μας είπε ότι θα επανέλθει στο ζήτημα του σκρουμπιού. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αποθετηθώ για το είδος αυτό. Και στη συνέχεια Έχουμε το ζήτημα της κυρίας Άντρας Περέας όσον αφορά την κατάρτιση και όσον αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Με την εμπειρία που έχουμε πλέον τα τελευταία τρία χρόνια και στο συντονισμό που έχουμε πετύχει για τον έλεγχο της αλίας ερυθρού τόνου, ένας εκπρόσωπος κράτους μέλους πριν από μερικές εβδομάδες μου είπε η βασικότερη συμβολή της υπηρεσίας μας είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γιατί στο παρελθόν υπήρχε πολύ μεγάλη απουσία εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία. Μου είπε λοιπόν η συναδελφή μου αυτή ότι η βασική συμβολή μας είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη γιατί καταλαβαίνετε ότι ε, αυτές οι επιχειρήσεις επιτήρησης γίνονται από κοινού, από πολλά κράτη-μέλη. Ο συντονισμός επιτυγχάνεται από κοινού μέσω της υπηρεσίας μας και εφαρμόζεται από κοινού επιτόπου. Η όλη διαδικασία λοιπόν πλέον είναι συλλογική, είναι πολύ πιο διαφανής και αυτό έχει οδηγήσει σε ένα πολύ καλό κλίμα εμπιστοσύνη να στα κράτη-μέλη. Και αυτό με τη σειρά του διευκολύνει την επιβολή των κανόνων της κοινή ελευτικής πολιτικής και τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και για τους ίδιους τους αλείς. Είναι σε θέση πλέον να δούνε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουμε εμεί μια διακριτική μεταχείριση ανάμεσα στο είδος του σκάφους ή στην εθνικότητα των αλλιέων. Οι επιτηρήσει είναι κοινέ και για όλους, δεν επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά γίνονται σε όλες τις γεωγραφικές εκείνες ζώνες όπου παρατηρείται ελευτική δραστηριότητα. Γιατί ξέρετε πολλές φορές ε, παραπονιούνται από τον αλευτικό τομέα ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στις ε, επιτηρήσεις μας. Τουλάχιστον όμως δεν ε, καταγγέλουν μεροληπτική εφαρμογή των κανόνων ή των επιτηρήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία και πιστεύω ότι έχουμε όντως συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη να είμαστε στα κράτη-μέλη. Και το ζήτημα της κατάρτισης βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, η κατάρτιση για τους επιτηρητές. Αυτή είναι ένα σημαντικό δίδαγμα που έχουμε από το όλο εγχείρημα για τον ρηθρό τόνο. Για παράδειγμα, η Ιταλική ακτοφυλακή έχει 9.000 προσωπικό. Θεωρητικά θα μπορούσαν όλοι να κάνουν επιτήρηση. Ένα μεγάλο τμήμα όμως αυτών των 9.000 υπαλλήλων δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια σαρδέλα και σε έναν ερυθρό τόνο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει κατάρτιση, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλά εξειδικευμένη και κατηρτισμένη ομάδα ε, ελεγκτών, επιτηρητών που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την επιτήρηση. Αυτό προσπαθούμε ακριβώς να κάνουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καλά κατηρτισμένες ομάδες οι οποίες μπορούν έπειτα να αναπτύσσονται σε ε, ετήσια βάση σε διάφορες περιοχές. Νομίζω ότι μίλησα για τις παραβάσεις. Το είδος των παραβάσεων μπορείτε να το δείτε στον πίνακα αυτό. Μπορείτε να δείτε το σκάφος και από ποια χώρα προέρχεται. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα, για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τις ε, εκθέσεις που μας αποστήλατε. Θα ήθελα να παρακαλώ στους συναδέλφους να τις διαβάσουν εκθέσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες, κυρίως αυτή που αφορά την αλίευση του ερυθρού τόνου, διότι πρόκειται για μία έκθεση πολύ λεπτομερή. Και βεβαίως αύριο θα δούμε και το ντοκιμοντέρ αυτή της BBC. Είπατε ότι πρόκειται για δεδομένα πρώτερα του 2010 και έχουν γίνει μεγάλη πρόοδοι από τότε. Όπως πάντα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επισκεψή σας στην Επιτροπή Αλίας και για τις εκθέσεις και πάλι που όπως πάντα είναι πολύ αποσαφινιστικές και μας βοηθούν να καταλάβουμε τα προβλήματα. Bueno, con esto pasamos al siguiente punto. Και τώρα περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 6. Πρόκειται για μία ένα σημείο και κλεισμένο, που θα συζητήσουμε και κλεισμένο των θυρών. Παρακαλώ. Λοιπόν. Όλους όσους δεν έχουν δουλειά εδώ, υπαλλήλου, αξιωματούχους, να φύγουν από την έκθεση.